Λοιπόν, συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Σε ό,τι φορά τι αποφάσει των συντονιστών, φαντάζομαι καταλάβατε όλοι ότι η αναπουσία των συντονιστών αναβλήθηκε και η συνεδρία των συντονιστών. Οπότε περνάμε στην έκθεση για τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τη συντάκτρια της γνωμοδότησης μας, γιατί επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ακούσουμε λοιπόν την εισηγήτριά μας, την κυρία Κριστίν Ρεβό Νταλόν Μπονφουά. Έχεις το λόγο, Κριστίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση που σας προτείνω σέβεται τη λογική της Επιτροπής προτείνοντας ταυτόχρονα μία ενίσχυση των στόχων και ε, αποκαθιστώντας την αρχή του μπόνους μάλους. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την, παράμετρο της χρησιμότητας που απλώς περιπλέκει ε, την νομοθεσία ενθαρρύνοντας τα πιο βαριά και ρηπογόνα αυτοκίνητα. Θέλουμε περισσότερα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών ή χαμηλών εκπομπών και τεχνολογική ουδετερότητα, ώστε να ε, επιτρέψουμε στη βιομηχανία μα να παραμείνει ανταγωνιστική. Δηλαδή, οι ασιατικέ αυτοκινητοβιομηχανίε θα κυριαρχήσουν στο μέλλον στην αγορά μα με νέα οχήματα. Και οι δοκιμέ εκπομπών θα πρέπει να είναι πιο αυστηρέ, με ε, πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ε, αυτό θα πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι απλώς εργαστηριακές δοκιμές. Επίσης, ε, οι μετρήσεις μόνο στην εξάτμιση δεν επαρκούν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει μια μεθοδολογία υπολογισμού όλων των καυσέριων της διάρκειας ζωής του οχήματος που μπορεί να είναι χρήσιμη κατά την αναθεώρηση, η αναθεώρηση του κειμένου το 2024. Θα πρέπει επίσης να κρατήσουμε και ενδιάμεσους στόχους το 2025 έτσι μόνο η αυτοκίνητο βιομηχανία θα ανασκουμποθεί και θα μπει σε έναν ενάρετο κύκλο και μια προσπάθεια μείωση των εκπομπών. Η ΔΕΜΗ δεν θα έχουμε κανένα πρότυπο νέο για διοξείδιο του άνθρακα μεταξύ 2021 και 2030. Κάτι αδιανόητο εν ώψη τη επιτακτική ανάγκη να καταπολεμήσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ. Βέβαια, κάτι τέτοιο προποθέτει μια ρηξικέλευτη αλλαγή του βιομηχανικού μα μοντέλου, που δεν θα είναι ούτε απλή, ούτε εύκολη. Ε, η προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή, αλλά για να στεφθεί με επιτυχία θα πρέπει να είναι συνεπής με τη στρατηγική για τα εναλλακτικά καύσιμα και το σχέδιο για τις... αναμένεται το Μάιο ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μπαταρίες. Επίσης, ε, με τη νέα κινητικότητα μιλούμε για νέες θέσει απασχόληση, αλλά δύσκολη θα είναι η κατάσταση στα εργοστάσια αλλά ήδη έχουμε τη νέα κινητικότητα, οπότε θα πρέπει να είμαστε προορατικοί και διορατικοί για να μην αφήσουμε κανέναν στην άκρη, εξασφαλίζοντας φυσικά και την ανταγωνιστικότητά μας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Αυτά και περιμένουμε ανυπομονησία τους και συγγετές. Σας ευχαριστώ. Οποία λακωνικό της λαμπρά κυρία εισηγητρία. Α, θα ακούσουμε το τον κύριο Σαλίνη, το σκιώδη συγγετή από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω την τύχη να είμαι εισηγητής για το ΕΛΚ στο θέμα αυτό και στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Επιτροπή Ήτρε. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία επί των οποίων θα πρέπει να βρούμε κάποια κοινά σημεία διότι δεν έχουμε απόλυτη ταύτιση απόψεων με την συντάκτρια της γνωμοδότησης. Βέβαια, βλέποντας και όσα είδα στη συζήτηση στην Επιτροπή Ήτρε, υπάρχουν κάποια καθησυχαστικά στοιχεία στην πρόταση της ε, συντάκτριας. Καταρχάς, ε, αντιμετωπίζει σωστά κατά την άποψή μας το θέμα της ε, τεχνολογικής ουδετερότητας. Ιδιαίτερα νομίζω ότι είναι πολύ συνεκτικό και σέβεται πιστά το κριτήριο της ε, τεχνολογικής ουδετερότητας η πρόταση για τον συντελεστή διόρθωσης, ε, στον οποίο λαμβάνεται υπόψη με σωστό τρόπο και η συμβολή των εναλλακτικών καυσίμων για την επίτευξη των γενικών στόχων που έχουν καθοριστεί από το Παρίσι και των πιο συγκεκριμένων που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα τα θέματα τα οποία αφορούν την αναθεώρηση των στόχων, δηλαδή τον ενδιάμεσο στόχο που υπενθυμίζεται εδώ ε, και που η Επιτροπή προτείνει να είναι στο 15% μέχρι το 2025 και το 2030 η πρόταση είναι για 30%. Το ε, αρχικό ε, ποσοστό που προτείνει η συγγήτρια μου φαίνεται λίγο υπερβολικό και εδώ νομίζω ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να πιέσουμε ε, υπερβολικά το σύστημα ε, και έτσι θα έχουμε και ε, στρέβλωση ακόμα και στην ίδια τη βιομηχανική παραγωγή. Κάτι το οποίο θα έχει ως συνέπεια να μην δώσουμε τη δυνατότητα να επιτευθούν οι στόχοι που προβλέπονται από το Παρίσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όπως είναι γνωστό, το 2017 η αγορά αυτοκινήτων diesel είχε μια πτώση πάνω από το 4%. Αλλά η αγορά οχημάτων ε, που ε, κινούνται με βενζίνη αυξήθηκε κατά 10%. Το αποτέλεσμα είναι ότι ε, ρηπαίνουμε περισσότερο το περιβάλλον. Επομένως, οι διαδικασίες αλλαγής ακόμα και όταν ή μάλλον κυρίως όταν ο στόχο που θέλουμε να πετύχουμε είναι απόλυτα σωστός, θα πρέπει ε, να ε, γίνονται με ρεαλισμό και σαφήνεια, διότι το να καταστρέψουμε ένα βιομηχανικό σύστημα με στόχους που είναι αδύνατο να επιτευθούν, έχει ε, σαν συνέπεια ότι ε, ζημιώνουμε μόνο την κοινωνία των πολιτών. αυτό λοιπόν το οποίο προτείνουμε και είναι το σωστό, είναι να επιτρέψουμε στον νομοθέτη να εγγυηθεί στους πολίτες να επιτευχθούν τα σωστά αποτελέσματα που έχουμε καθορίσει στο Παρίσι. Ιδάλλως θα υπάρχει μία γραμμή παραγωγής. Σκεφτείτε όλους τους ε, μικρούς ε, προμηθευτές ε, της αυτοκινητοβιομηχανίας που μέσα σε λίγα χρόνια θα πρέπει να θα βρεθούν με προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να πουληθούν πουθενά στην αγορά. Εν τω μεταξύ, ο καταναλωτή δεν θα δέχεται αυτή την πρόκληση, διότι όπω είπα προηγουμένω, ο καταναλωτή θα ψάξει ούτω ή άλλω να βρει το φθηνότερο αυτοκίνητο. Επομένω, σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο πρέπει να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε συνέπεια και ισορροπία και φυσικά το σημείο κίνηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα επιτρέπει να το επιτύχουμε αυτό και θα ήθελα να προτείνω στου συναδέλφου να ξαναδούν όσο το δίνουν περισσότερο τις απαιτήσει μας, που μπορεί να είναι και ιδανικές για έναν τέλειο κόσμο, και να προσπαθήσουμε εδώ, σε αυτή τη διαδικασία, να έχουμε μια πραγματικά βιώσιμη διαδικασία ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Σαλίνη. Για το ECR, το λόγο έχει ο κύριος Τωσανόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι η προσέγγιση της συντάκτρια γνωμοδότης είναι ρεαλιστική, επικοδομητική και πολύ θετική. Μου αρέσει ιδιαίτερος. Θα πρέπει ε, να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί και να μην πιέσουμε υπερβολικά την αυτοκινητοβιομηχανία και την οικονομία. Επίσης, πρέπει να είμαστε αυστηροί και να ενισχύσουμε κάποια κριτήρια. Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διοξίδιο του άνθρακα, θεωρώ ότι η πρόταση συγκήτριας είναι η καλύτερη βάση για τη συζήτηση. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε πολύ θετικές συμβαστικές προτάσεις, γιατί σε μεγάλο βαθμό Συμφωνώ με την εισηγητρία για την ανάγκη τεχνολογικής ουδετερότητας. Αυτό το σημείο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλαχθεί. Όταν ε, οι πολιτικοί περιορίζουν υπερβολικά και οριθετούν υπερβολικά την κατεύθυνση της τεχνολογίας, ε, τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά. Γι' αυτό η προσέγγιση της ε, ουδέτερη τεχνολογικά μεθόδου είναι η καλύτερη. Παρόλο που υπάρχουν και άλλα συστήματα, έχουμε καύσιμα από υδρογόνο, από φυσικό αέριο, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν ξέρουμε από τώρα με βεβαιότητα προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί ο κόσμος. Μπορεί στο μεταξύ να προταθούν νέες καινοτόμες λύσεις μπορεί να γίνουν κάποιες, κάποιες ρηξικέλευθες εφευρέσεις για τις μπαταρίες, για παράδειγμα. Και αυτό ίσως θα αλλάξει το τοπίο. Ας μην οριθετήσουμε υπερβολικά λοιπόν την τεχνολογία. Τεχνολογικά ουδέτερη πρόταση. Τώρα, για τον οργανισμό που θα διενεργήσει την εποπτεία, την επιτήρηση. Και αυτό το σημείο θα πρέπει να συζητηθεί προσεκτικά και διεξοδικότητα για να αποφύγουμε υπερβολική γραφειοκρατία και διοικητικό άχθος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Γενικώ η πρόταση μου φαίνεται ρεαλιστική, ορθολογική και τα υπόλοιπα θέματα θα τα αντιμετωπίσουμε με τροπολογίες. Γενικώ πάντως η έκθεση είναι καλή και συγχαρητήρια στη συντάκτρια της γνωμοδότησης. Ευχαριστούμε κύριε Τωσενόφσκι. Για τους φιλελεύθερους το λόγο έχει ο κύριος Ράντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και οι οδικές μεταφορές, 20% όλων των εκπομπών ε, θερμοκηπίου του άνθρακα, ε, σίγουρα ε, μάλιστα τα, τα νέα γιοταχή τα και τα ημιοφορτηγά είναι ε, πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό ρήπανσης με καυσαέρια στις οδικές μεταφορές, οπότε είναι λογικό να αντιμετωπίσουμε με τέτοιες προτάσεις αυτά τα προβλήματα. Συμφωνώ με τη συντάκτρια της γνωμοδότησης και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να χορηγήσουν αξιόπιστες ε, πληροφορίες και ε, η συγκέντρωση των στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει με βάση συνθήκε πραγματική οδήγηση και όχι εργαστηριακέ δοκιμέ. Επίση, ε, συμφωνώ και εγώ, ε, δεν θα πρέπει με αυστηρές, αυστηρούς στόχους για τα αέρα του θερμοκηπίου δεν θα πρέπει να τιμωρήσουμε κάποια οχήματα μηδενικών εκπομπών. Επίσης να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, καυσίμων νέας γενιάς που θα έχουν λιγότερες εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου. Συμφωνώ λοιπόν με τις σχετικές προτάσεις της κυρίας Ρεβόνταλόν να συμπεριληφθούν και αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα στην οδηγία και να τα εντάξουμε πολύ καλύτερα στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που δεν το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σωστό τρόπο. Γι' αυτό και οι δικές μας τροπολογίες αυτή την κατεύθυνση θα έχουν, να συνδυάσουν δηλαδή τις δύο αυτές οδηγίες και α, κανονισμούς, ώστε να έχουμε ένα ενιαίο πακέτο. Σε ό,τι αφορά ε, την πρόταση το 2040, όλα τα νέα οχήματα να είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών, παρά είναι φιλόδοξη η πρόταση. Και επίσης η μείωση των εκπομπών κατά 15% μέχρι το 2025, ε, σε 20% για τα ημιφορτηγά και 25% για τα ιοταχή, ενώ για το 2030 30%, από 30% να είναι 40% και 50%. Ε, οι φιλελεύθεροι είναι ανοιχτοί να συζητήσουν αυτές τις ε, προτάσεις για τα διαφορετικά ποσοστά σε ό,τι αφορά τα καυσαέρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταλούντα εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, την εισηγήτρια για μια εξαιρετική γνωμοδότηση. Μιλώ εκ μέρου του συναδέλφου που δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει ε, στα καθαρά αυτοκίνητα για να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματος, ε, αλλά ε, και για να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα ε, και έχουμε καθυστερήσει ε, σε σχέση με την Καλιφόρνια, την Κίνα και την Ιαπωνία όσον αφορά την ηλεκτροκινητικότητα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ανεπαρκής. Χρειαζόμαστε πιο υψηλούς στόχους, πιο φιλόδοξους και συμβατούς με τη Συμφωνία του Παρισιού. Για ε, το νέο στόλο αυτοκινήτων ε, μέχρι το 2025 στόχο 45% και 75% για το 2030 λέει, ε, είναι η πρότασή μας, η οποία μπορεί με την πρώτη ματιά να φαίνεται υπερβολική, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό έχει να κάνει με τις πωλήσει νέων αυτοκινήτων, όχι με τον υπάρχοντα στόλο. Αυτό είναι φιλόδοξο, είναι όμως εφικτό. Μάλιστα η Volvo σκοπεύει μέχρι το 2025 ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν το 50% των πολίσεων του σε κάτι που ευθυγραμμίζεται με τις δικές μας ε, πράσινε ε, προτάσεις. Ε, πρέπει να ενθαρρύνουμε την παραγωγή αυτή. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις στην αγορά όσον αφορά ε, ε, τις δυνατότητες φόρτισης ε, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την ομαλή μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Χρειάζεται λοιπόν υποδομή φόρτιση των αυτοκινήτων αυτών για να ενθαρρύνουμε την πώληση αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Θα πρέπει να επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, τους νέους τρόπους κατασκευής και τις νέες δεξιότητες. Ε, πιστεύω ότι ε, θα μπορέσουμε να έχουμε ομαλή μετάβαση όσον αφορά τον στόλο αυτοκινήτων μας ε, εάν δώσουμε τα απαραίτητα κίνητρα, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και στην εξαγωγή καθαρών αυτοκινήτων στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταλίντε. Η κυρία Κίλονεν από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω ε, την ε, εισηγήτρια. Έχει συνδυάσει με έξυπνο τρόπο διάφορα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η δουλειά που έχει κάνει. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και τις τεχνολογίες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τη σχέση με τα καύσιμα. Εμένα θα με ενδιαφέρε να εξετάσουμε περαιτέρω ε, τον κύκλο ζωής των διαφόρων αυτοκινήτων, των διαφόρων είδων οχημάτων διότι τώρα εξετάζουμε μόνο τις εκπομπές όταν ε, βρίσκονται σε χρήση. Επίσης, ε, ο κύκλος ζωής των συστημάτων ενέργειας και του συνόλου του οχήματος. Τι, πόση ενέργεια καταναλώνεται για την κατασκευή ενός οχήματος. από πού προέρχεται η ενέργεια αυτή. Με ενδιαφέρουν επίσης τα βιοκαύσιμα που παράγονται από απορρίμματα. Επίσης τα νέα ε, παραφινικά καύσιμα που ε, είναι η καινοτομία στον τομέα των βιοκαυσίμων. Δεν θέλω να εξετάζουμε απλά μία τεχνολογία και μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Με ενδιαφέρει γενικότερα ο κύκλος ζωής των οχημάτων, οι διάφορες λύσεις και οι διάφορες τεχνολογίες που υπάρχουν, διότι είναι επίγουσα η ανάγκη να έχουμε ένα ευρύτερο καλάθι επιλογών και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πολύ καλή δουλειά πάντως και προσλέπω στην συνέχιση της συνεργασίας με την εισηγήτρια και τους Θα Σας ευχαριστώ κυρία Κίλωνεν. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους ευρωβουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο, ο κύριος Κόχ. Κυρία εισηγήτρια, αγαπητή Κριστίν, σε ευχαριστώ ευχαριστώ για την εξαιρετική σου έκθεση που όμως σε κάποια σημεία μου φαίνεται ότι υπερβάλλει. Δεν χρειαζόμαστε ε, ευρωπαϊκό οργανισμό για την εποπτεία της αγοράς ε, της ε, οδικής κυκλοφορίας. Το Συμβούλιο συμφώνησε να μην δημιουργήσει ένα τέτοιο οργανισμό. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, να γίνουμε ρεζίλια επανερχόμενοι στο ζήτημα αυτό. Συνεχίζω επίσης ε, να είμαι τη άποψη ότι ο στόχο για το 2030 αρκεί. Δεν χρειαζόμαστε ενδιάμεσο στόχο για το 2025. Είμαι πεπισμένο γι' αυτό, όχι μόνο επειδή χρειαζόμαστε ασφάλεια προγραμματισμού στη βιομηχανία, αλλά επειδή πρέπει να θέτουμε φιλόδοξου ε, και επιτεύξιμου στόχου. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη ακόμα περισσότερο πέρα από, τις, ε, από τους ήδη φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ε, φυσικά, ε, φυσικά τα οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών είναι το μέλλον. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και το οικολογικό αποτύπωμα των καυσίμων και δεν ε, θα πρέπει απλά να θεωρούμε ότι ο διάβολος ε, είναι οι, μηχανές οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Συνεχίζω να πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ουδέτεροι ως προς την τεχνολογία στις προτάσεις μας. και δεν ε, μπορώ να συμφωνήσω με, υπολογισμό, με επανυπολογισμό των ε, εκπομπών. Και νομίζω ότι ήδη αυτά που έχουμε στα χέρια μας είναι αρκετά καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόχο. Κύριος Πίπερ. ευχαριστώ πολύ. Δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Ε, συμφωνώ με όλα όσα είπε ο συναδερφός Κόχ όσον αφορά τον ε, νέο οργανισμό. Συμφωνώ απολύτω. Βέβαια, αν, ε, ε, ε, εάν δημιουργηθεί στην δική μου εκλογική περιφέρεια, τότε θα τον στήριζα. Αλλά κατά τα άλλα συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Κόχ. Όσον αφορά την Volvo, όπως ανέφεραν οι πράσινοι, η Volvo είναι εταιρεία χωρίς ούτε ένα οικολογικό όχημα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να την αναφέρουμε ως ε, υπόδειγμα. Όσον αφορά την έκθεση και ε, τις ε, ενέργειες στις οποίες θέλετε να επιβάλλετε κυρώσεις, νομίζω ότι είναι υπερβολική έκθεση στο θέμα αυτό. Εάν θέλουμε να κινηθούμε προς την ηλεκτροκινητικότητα, αυτό στη Γερμανία θα σημαίνει το εξής. Ε, έχουμε μεν ε, ηλεκτρικά οχήματα, αλλά κατά 45% τα, η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τα οχήματα αυτά προέρχεται από ε, λιγνητικές μονάδες. Θα πρέπει λοιπόν όσον αφορά τους στόχους αυτούς, ε, να εξετάζουμε μαζί τα πράγματα αυτά. Δηλαδή, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, θα πρέπει να συνοδεύει αυτά που αναφέρουμε εδώ πέρα. Διότι αλλιώς θα πετύχουμε το αντίθετο από αυτό που θέλουμε να πετύχουμε από περιβαλλοντικής πλευράς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίπερ. Η κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Πιστεύω ότι είναι πολύ λογικό να προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα για το 2030, το οποίο να συνάδει με τους γενικούς στόχους της Ευρώπης όταν αναφερόμαστε σε μείωση εκπομπών. Επιπλέον, ε, είμαι πεπισμένη ότι το επίπεδο φιλοδοξίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τη συμπεριφορά των πολιτών όταν αγοράζουν οχήματα. Επομένως, ε, να έχουμε κατά νου ότι οι ευρωπαϊκές αγορές ε, είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη θα υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε ένα σύστημα για να παρέχουμε σημαντικά κίνητρα, ενώ σε κάποια άλλη, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, δεν φαίνεται να πληρούνται οι προποθέσει για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν, κατά την άποψή μου, στο ενδιάμεσο τη πορεία να μπορέσουμε να κάνουμε μια αξιολόγηση με ένα σαφέ πλαίσιο όσον αφορά τη χρήση οχημάτων ε, που τροφοδοτούνται ε, με εναλλακτικά καύσιμα και εν ώψη της αλλαγής της τεχνολογίας και για τα οχήματα τα οποία θα είναι παρόντα στους ε, δρόμους μας να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια περαιτέρω ε, πιο φιλόδοξα αποτελέσματα. Τέλος, μια παρατήρηση που αφορά τη σύγκριση μεταξύ ε, φορτηγών για μεταφορά εμπορευμάτων και αντιστρόφως οχημάτων επιβατικών. Διότι ε, θεωρώ ότι πρόκειται για τελείως διαφορετικούς τομείς ε, και επομένως ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και ανάλογη διαφοροποίηση για τα θέματα αυτά στον τομέα και να το εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντεμόντε. Ο κύριος Κράμερ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Ο κύριος Ράντος είπε ότι ε, οι ε, μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 30% των εκπομπών ε, και τις έχουμε αγνοήσει τελείως, δεν τις έχουμε συμπεριλάβει στον υπολογισμό και γι' αυτό δεν τις υπολογίζουμε. Πριν 30 χρόνια στη Γερμανία αποφασίσαμε να ε, έχουμε χαμηλή φορολογία στο ντίζελ και έτσι έχουμε ακόμα αρνητικό ισολογισμό στις ε, εκπομπές και πρόσφατα οι ομοσπονδιακές αρχές είπαν ότι έχουμε 6.000 πρόωρους θανάτους το χρόνο λόγω των ε, εκπομπών οξυδίων του αζότου. 6.000 προώρους θανάτους έχουμε στη Γερμανία λόγω του ντίζελ. Αυτό όμως δεν έχει αλλάξει την επιδότηση του ντίζελ. Ενώ οι σιδηροδρομικές εταιρείες ε, εποφελούνται από το ντίζελ, ε, δεν ε, κάνουν κάτι διότι ανταγωνίζονται τις οδικές μεταφορές. Τώρα λοιπόν ε, μιλάμε για τις ε, μπαταρίες των αυτοκινήτων, για τα φωτοβολταϊκά. Θα πρέπει να εξετάσουμε συνολικά την παραγωγή, την χρήση και κυρίως την ανακύκλωση των οχημάτων αυτών. Να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση και να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη λύση με βάση τον συνολικό κύκλο ζωής. Και ο κύριος Πίπερ έχει δίκιο. Στην ε, Γερμανία είμαστε ε, περήφανοι για τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όταν έχουμε ηλεκτροκινητικότητα, από πού προέρχεται η ενέργεια. Από ε, μονάδες παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη, από θερμοηλεκτρικά εργοστάσια και Αυτά μολύνουν πολύ το περιβάλλον. Χρειάζεται λοιπόν μια γενικότερη οπτική. τέλο στον Τίτερ Κοχ να πω ότι 2030, όχι 2025, γνωρίζετε του στόχου. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι πάντα είναι ωραίοι. Αλλά εάν δεν κάνουμε το πρώτο βήμα, τότε δεν θα πετύχουμε ούτε το δεύτερο ούτε το τρίτο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και βραχυπρόθεσμου στόχου. Μπορούμε να συζητήσουμε το ύψο του, αλλά το να λέμε ότι θα έχουμε 12 χρόνια περιθώριο και στο μεταξύ η αυτοκινητοβιομηχανία απλά να κλέβει τον χρόνο αυτόν ε, δεν έχει κανένα νόημα. Στο μεταξύ δηλαδή δεν θα κατηγορηθεί κανένας, ε, δεν θα γίνουν ε, έρευνας, θα έπρεπε να έχουμε μάθει από το Dieselgate. Γι' αυτό χρειαζόμαστε βραχυπρόθεσμους στόχους για να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Και εγώ θα ήθελα λίγο το λόγο για να κάνω κάποιες σκέψεις. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι παρά την ε, βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων τα τελευταία 15 χρόνια ε, των οχημάτων, γιατί έχουμε λιγότερα καυσαέρια, έχουμε καλύτερο έλεγχο των καυσαερίων των οχημάτων, παρόλα αυτά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω της αύξησης του όγκου ε, της κυκλοφορίας των οχημάτων. Και υπάρχουν πολλοί παράγοντες ε, που οδηγούν στην επιδείνωση. Σίγουρα η μεικτή συνολική επίδοση των οχημάτων είναι το ένα στοιχείο, αλλά υπάρχουν και κάποια κοινωνικά και συμπεριφορολογικά προβλήματα. Βέβαια μπορεί να μην είναι του παρόντος, αλλά επηρεάζουν την κατάσταση. Οι εκπομπές ενός αυτοκινήτου που έχει 80 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα το χιλιόμετρο, δεν είναι το ίδιο αν είναι ένας ε, μόνο επιβάτης ή πέντε. Εμένα με ενδιαφέρει πόσο και πώς ε, κάνουμε τις μεταφορές. Θα πρέπει να υπάρχει και κοινωνική παράμετρος, ε, ε γιατί επηρεάζει τις εκπομπές ε, ανά χιλιόμετρο. Είναι σημαντική αυτή η παράμετρη. Γιατί όταν οδηγώ μόνος μου δεν παραγωγώ τόσα καυσαέρια όταν έχω ε, πέντε επιβάτες, συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο. Επίσης, ε, έγινε επανάληψη της χθεσινής συζήτησης που είχαμε στην Ήτρε. Τρεις ε, είναι συγκρουμένοι στόχοι και περιλαμβάνονται στον ίδιο κανονισμό. Υπάρχει ο, περι, ο περιβαλλοντικός στόχος, ο τεχνολογικός και ο οικονομικός στόχος. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ του. Και όσο πιέζουμε προς τον ένα στόχο, ε, χρειάζεται να βλύνουμε τον άλλο στόχο. Όταν πιέζουμε στον περιβαλλοντικό στόχο, θα αυξηθεί ο οικονομικός κίνδυνος. Ε, γιατί όσο πιο αυστηρίες είναι οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές, τόσο πιο δύσκολα θα ακολουθήσει η αυτοκινητοβιομηχανία. Ε, βέβαια, αν εξαρτάται από την αυτοκινητοβιομηχανία, δεν θα γινόταν αλλαγές. Είναι δύσκολο να συμβιβάσουμε όλους αυτούς τους στόχου που μερικές φορές είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Άλλοι έχουν μεγαλύτερες περιβαλλοντικές ευαισθησίε, άλλοι περισσότερο οικονομικές ευαισθησίε. Τρίτο σχόλιο. Να δούμε και την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είμαι φανατικός οπαδό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αλλά ε, πρόκειται για μια συνέχεια στην προσέγγιση με κανονισμό που τροποποιεί προηγούμενο. Είμαστε έτοιμοι για κάποιες κανονιστικές τομές όπως πρότεινε Αμερική. Μερικές φορές διπλασιάζοντας τις προτάσεις. Εκεί που υπολογίζουμε με γραμμάρια να περάσουμε από το 30% στο 75% αυτό πραγματικά είναι μια πρόταση που φέρνει ρήξη. Η παρούσα κατάσταση δικαιολογεί μια τέτοια στάση ρήξης. Γιατί αναμένονται τεχνολογικές βέβαια εξελίξεις που λένε ότι θα μας επιτρέψουν τέτοια μεγάλη φιλοδοξία. Πριν από 7-8 χρόνια μας ε, παρουσίαζαν ε, την κατάσταση ότι από το 2015 θα είχαμε αστρονομική αύξηση των ηλεκτρικών ε, αυτοκινήτων. Κάτι που δεν έγινε. Οπότε προσοχή στις προβλέψεις. Προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Επίσης όλοι επέμειναν στην ε, ε, τεχνολογική ουδετερότητα και νομίζω ότι πολύ σωστά το έκαναν. Ούτε από ποσοτική ούτε από ποσοτική άποψη έχουμε την πολυτέλεια κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να μείνουμε τεχνολογικά ουδέτεροι. Επίσης και η αιρεσιμότητα είναι τμήμα του σεβασμού της τεχνολογικής ουδετερότητας. Γιατί δεν μπορούμε μια μόνο κοντιλιά να διαγράψουμε την αιρεσιμότητα από τους κανονισμούς, γιατί είναι σημαντικό στοιχείο της οικονομικής διάρθρωσης. Δεν λέω ότι θα πρέπει να την υπερασπίσουμε κάθε πάση θυσία την αιρεσιμότητα, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο άκαμπτοι και αδιάλακτοι. Μιλήσαμε για το συνολικό ισοζύγιο, συμφωνώ και για τον οργανισμό. Και εγώ είμαι υπέρμαχος του οργανισμού. Ούτως ή άλλως έχει υπερψηφιστεί στην ε, Επιτροπή εμείς. Και ε, οριακά κατέπεσε στην Ολομέλεια. Οπότε θα πρέπει να απελπιζόμαστε. Δεν αποκλείεται να γίνει τελικά. Και τέλος, το θέμα των υποδομών αναφέρθηκε από κάποιους συναδέλφους. Οι υποδομές που θα επιτρέψουν στα νέα οχήματα να γεμίζουν το τεπόζιτό τους με τα νέα καύσιμα. Πάντως, όταν αλλάξει η αυτονομία των οχημάτων, και μιλάω για τα ηλεκτρικά, θα αλλάξει τελείως και το ζήτημα των υποδομών. Και αν στην πρώτη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουμε αυτονομία 120 χιλιόμετρα, που ήταν ο μέσος όρος, τώρα θα πρέπει να βρούμε ε, κάθε 100 μέτρα ουσιαστικά να φορτώνουμε στα, στο οδικό δίκτυο. Αν όμως η αυτονομία είναι 500 χιλιόμετρα, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πού θα συγκεντρώσουμε τις ε, υποδομές για γρήγορη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκίνητων. Οπότε, πολύ σύντομα θα φτάσουμε στα οχήματα και τρίτης ε, γενιάς. Τώρα είμαστε στη δεύτερη γενιάς ηλεκτρικά οχήματα. Και σίγουρα ο καθένας θα προωθεί τις δικές του προτεραιότητες. Καλύτερα να μείνουμε σε ορθολογικές λύσεις. Ορθολογική ε, ε ουδετερότητα τεχνολογική, αναφέρθηκαν τα 13 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, προσοχή να μην επηρεάσουμε το μέλλον. μπορούμε να αφανίσουμε την βιομηχανία αν την περιορίσουμε υπερβολικά. Ισμαήλ Ερτούκ, και εσύ αν δεν κάνω λάθος ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω το θέμα εδώ δεν είναι τα αγαπημένα θέματα του καθενός, αλλά η τεχνολογική ουδετερότητα. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και στο μέλλον την τεχνολογική ουδετερότητα. Δεύτερον, πολλά υπόθηκαν. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα λογικά. Ο συνάδελφος Κράμερ μίλησε για τις στατιστικές ε, για ε, τους πρόορους θανάτους. Ε, αυτό μια στατιστική είναι. Ο κύριος Πίπερ μίλησε για το 45% του ηλεκτρικού ρεύματος που προέρχεται από θερμοηλεκτρικές μονάδες. Εάν δίνουμε κίνητρα ε, για την ηλεκτροκινητικότητα ε, και την πράσινη τεχνολογία, τότε θα μειωθεί το ποσοστό ε, της θερμοελεκτρικής ενέργειας και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν το αγαπημένο θέμα του καθενός είναι το περιβάλλον ή η κινητικότητα. Το βασικό θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η βιομηχανία στην Ευρώπη, ιδιαίτερα η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, θέλουμε να είναι κορυφαία σε 20, 25, 30 χρόνια. Καλές προθέσεις έχουμε, μπορεί κανείς να δώσει τα παραδείγματα της Κόντακ, ε, της Nokia κλπ. Εάν όμως έχουμε καλές προθέσεις απέναντι στη βιομηχανία μας, θα πρέπει να τις δώσουμε τη δυνατότητα να πετύχει τους στόχους που θέτουμε σε πολιτικό επίπεδο. Και οι στόχοι αυτοί δεν θα είναι χρήσιμοι για τη συνολική βιομηχανική ανάπτυξη αν είναι υπερβολικά επικής. Ούτε όμως και θα πρέπει να τους θέσουμε τόσο ψηλά ώστε να μην ε, μπορούν να επιτευχθούν μόνο και μόνο για να χαϊδέψουμε το πολιτικό μας εγώ. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας κατά νου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σωστά κατά τη γνώμη μου, έχει ε, θέσει και έναν ενδιάμεσο στόχο. Εάν δεν τον έχουμε αυτόν, τότε και η σχετική βιομηχανία δεν ε, θα πάρει σοβαρά το θέμα. η οδηγία για την υποδομή εναλλακτικών ε, καυσίμων θα μας είχε δώσει σήμερα ε, πολλές ε, δυνατότητες εναλλακτικές, αλλά με δικαιολογία τα εθνικά σχέδια χάσαμε πολύ χρόνο. Νομίζω θα μπορέσουμε να πετύχουμε φιλόδοξους στόχους και ήδη σήμερα θα πρέπει να προετοιμάσουμε τη βιομηχανία μας. ώστε να αποφασίσει εάν ε, θα πρέπει να καταργήσει βαθμιαία της, ε, την τεχνολογία εσωτερικής, εσωτερικής καύσης. Ε, εγώ δεν είμαι και βέβαιος ε, γιατί τίποτα. Δεν γνωρίζουμε τι θα μας φέρει το μέλλον, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε τεχνολογικά ε, ουδέτεροι. Θα πρέπει να εξετάσουμε μήπω ε, και με την τεχνολογία εσωτερική καύση μπορέσουμε να έχουμε τόσο χαμηλές εκπομπέ και όχι να θεωρούμε ότι από μόνη τη είναι κακή η τεχνολογία αυτή. Όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος ποντάρει στην ηλεκτροκινητικότητα, στην τεχνολογία του υδρογόνου, μπορεί να αγοράζουμε τα οχήματά μας αλλού και ε, να... και να έχει χαθεί όλη η βιομηχανία μας. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε η πιο ισχυρή οικονομική δύναμη στον κόσμο. Και η Κίνα με τα 1,3 εκατομμύρια πληθυσμό μπορεί να επιβάλλει μέτρα ε, και η Κίνα έχει υψηλό ποσοστό παραγωγής των οχημάτων αυτών. Εμείς όμως έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά πολίσεων. Ε, εμείς λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε τα οχήματα αυτά στους δρόμους μας. Νομίζω λοιπόν ότι καλά θα κάνουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα ώστε να προχωρήσουμε σε μια στρατηγική μείωση των εκπομπών ε, και να προσεγγίσουμε το θέμα με τρόπο τεχνολογικά ουδέτερο. Ευχαριστώ Ισμαήλ. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Θα μπορούσατε επί τη ευκαιρία να περιοριστείτε στα πέντε λεπτά εντό εισαγωγικών, γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όταν μιλά κάποιος για οχήματα, δύσκολα μπορεί να περιοριστεί στα πέντε λεπτά. Είναι τόσο σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πράγματι εξετάζει τρεις διαφορετικούς στόχους. Ο ένας είναι ο περιβαλλοντικός, ο δεύτερος είναι τι σημαίνει για τους καταναλωτές και τους πολίτες της Ευρώπης και το τρίτο είναι ο αντίκτυπος για την απασχόληση, η οποία φυσικά σχετίζεται στενά με την καινοτομία στο μέλλον. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα αναφέρθηκαν εδώ σήμερα το απόγευμα. Όσον αφορά τον περιβαλλοντικό στόχο, η πρόταση αυτή ε, υπάρχει προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να τηρήσει τη δέσμευσή τη ε, στη Συνθήκη των Παρισίων. Δηλαδή, μέχρι το 2030 ε, λιγότερες εκπομπές κατά 40%. Αν δείτε τις δεσμεύσεις μας, αυτό σημαίνει ότι οι οδικές μεταφορές θα πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον το 25% και αυτή η πρόταση από μόνη της θα επιτρέψει να φτάσουμε στο 22% μείωση. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που ε, υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μειώσουν ε, περαιτέρω τις εκπομπές ε, στα ποσοστά που χρειάζεται. Αυτό περιλαμβάνει τα καθαρά οχήματα, την, την ευρωβινιέτα, την οδηγία για τις μεταφορές και επίσης ε, οι εντολές ε, για το μείγμα των καυσίμων, ε, το blending και θα επανέλθω σε αυτό εντός ολίγου. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, την αποταμίευση για τους καταναλωτές, ο στόχος του 30% που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν ένα πλεονέκτημα το 2030, περίπου 1.400 ευρώ και αυτό φυσικά θα αποτελέσει κίνητρο για τους καταναλωτές για να αγοράζουν πιο καθαρά, λιγότερο ρηπογόνα δηλαδή οχήματα. Και αυτό φυσικά ε, σταδιακά θα υποχωρήσει, θα πέσει στα 400 ευρώ αν πάμε στο 40% και κατά 1000 ευρώ ε, αν πάμε στο 50%. Όσον αφορά την απασχόληση, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θεωρεί ότι θα υπάρξει ομαλή μετάβαση στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι σαφές ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να έχει περισσότερη καινοτομία, ιδίω όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Αλλά αν δείτε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό γίνεται με έναν τρόπο που επιτρέπει να γίνει ομαλά η μετάβαση. Επομένως, δεν θα υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος για την απασχόληση στην Ευρώπη. Μπορεί να υπάρξει και μια ελαφρά αύξηση. Ωστόσο, Εάν αρχίσουμε να προχωράμε πολύ πιο γρήγορα τη μετάβαση, τότε ε, θα υπάρχει ε, ίσως και κάποιος αντίκτυπος ε, ε, για την απασχόληση και αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Κάτι στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η τροπολογία 43, η οποία συνδέει την πρόταση για τα οχήματα με την κατανάλωση ανανεώσιμων ενέργεια, πηγών ενέργειας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσει κανείς. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι κάτι το οποίο σου προσέφερε όφελος από την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα σου προσφέρει ένα δεύτερο όφελος ε, στην νομοθεσία για τα οχήματα. Και αυτό σημαίνει διπλή καταμέτρηση. Και αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν μπορούμε να προσθέσουμε τις μειώσεις δύο φορές. Δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε δηλαδή στην απαιτούμενη μείωση στον τομέα των μεταφορών. Εάν θέλουμε να έχουμε κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά πολύ ψηλότερο στόχο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η συνολική μείωση στον τομέα των μεταφορών θα ε, προσμετρηθεί όπως απαιτείται. Μετά γίνεται μια μακρά συζήτηση για τον τύπο των μετρήσεων που θα πρέπει να γίνουν. Ο κύκλος ζωής αναφέρθηκε, ε, τα καύσιμα αυτές και οι πραγματικές εκπομπές κατά την ε, πραγματική οδήγηση, αυτά είναι θέματα τα οποία θα έρθουν σύν το χρόνο. Η Ευρωεπιτροπή γνωρίζει βεβαίως ότι πρέπει να γίνει κάτι από αυτού και υπάρχει κάτι σχετικό, αλλά το να περάσουμε σε τελείως διαφορετικό κύκλο δοκιμών από αυτόν που έχουμε τώρα, ε, θα χρειαστεί χρόνο, αρκετά χρόνια. Ο νέος κύκλος δοκιμών, το WLTP, μας πήρε έξι χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε ε, πραγματικό ε, τεστ, μάλλον τεστ πραγματικών εκπομπών κατά την οδήγηση θα χρειαστούμε πολύ χρόνο. Επομένως πρέπει να δούμε επίσης και τι θα μπει στο αυτοκίνητο, πόσο γρήγορα ε, οδηγεί κανείς, προς τα ποια κατεύθυνση. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα από έναν κύκλο δοκιμών απλώς σε σταθερή θέση. Ε, να επιστήσω την προσοχή σας λοιπόν σε αυτές τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει, διότι ορισμένε εξ αυτών θεωρούμε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτές εντός του χρονοδιαγράμματος που ε, μας προσφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. 11 δευτερόλεπτα παραπάνω μίλησα μόνο. Ευχαριστούμε. Η συγκεκριά μας τώρα. Η Κριστίν Ρεβό Νταλόν. Για τελευταία λέξη. Μια λέξη μόνο. Καμιά δύο τουλάχιστον. Αλλά όχι πολλές σίγουρα. Ευχαριστώ θερμά τους και οδησηγητές και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για τις παρατηρήσεις τους. Διαπιστώνω μία σύγκληση μεταξύ μας ως προς την ανάγκη να στηρίξουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τήρηση των δεσμεύσεών μα που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίση, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μπορούμε να συνδυάσουμε την οικονομική με την οικολογική προσέγγιση. Δεν είναι αλληλοσυγκρόμενε ή αλληλοαποκλειόμενε η οικονομική με την οικολογική προσέγγιση. Σα ίσα, συνδυάζοντα τε, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε μια καλή βιομηχανία και να έχουμε μια ποιότητα ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντάξια των φιλοδοξιών μας γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά ταυτόχρονα και φιλόδοξοι και να δώσουμε μια όθηση στους στόχους μας που δεν είναι για το απότερο μέλλον, αλλά για το εγγύς μέλλον. Επίσης, ε, χαίρομαι που για την τεχνολογική ουδετερότητα υπάρχει συνένεση και για το θέμα του κύκλου ζωής. και στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες πτυχές, γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα ε, τύπος αυτοκινήτου που θα παράγουμε στο μέλλον, αλλά θα συνεχίσουμε ε, να επεξεργαζόμαστε αυτή την ιδέα του συνδυασμού, του μίξ, του μείγματος που προτείνεται και θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Σε ό,τι αφορά τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ε, αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου θύμισε τις συζητήση που είχαμε στην Διερευνητική Επιτροπή, την ΕΜΙΣ. Εκεί ε, χάθηκε πολλής χρόνος, αλλά είναι κρίμα να λέμε, ε, να επικαλούμαστε τη δυσκολία για να αναβάλουμε την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Ακόμη και αν στην αρχή εφαρμοστεί πειραματικά, αλλά θα πρέπει να γίνει μια αρχή. Και όπως είπα πολλοί και το θέμα του ελέγχου επίσης είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει ο έλεγχος να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός. Και γι' αυτό είμαι υπέρ της ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα θέματα υποπτίας. Ραντεβού με τους και ηγετές τον Ιούνιο. Θα προβλέψω όσες συναντήσεις χρειαστούν για να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη πρόταση που ευελπιστώ θα συγκεντρώσει ε, τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Ευχαριστούμε κύριε Ρεβονταλόν. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η 17 Μαΐου 6 το απόγευμα. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Την ειδική ομάδα για τον τουρισμό και τη δημόσια κρόαση. Οπότε δίνω τις κοιτάλεις στον αρμόδιο αντιπρόεδρο για τα θέματα αυτά. Köszöntöm Η Επιτροπή έχει καθυστερήσει λίγο, αλλά θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε την Task Force για τον τουρισμό για ένα θέμα ε, το οποίο συζητήσαμε πολύ με το τουριστικό κλάδο μετά από μία σειρά συναντήσεων και εδώ στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, αποφασίσαμε να προωθήσουμε αυτή την ε, ε, πρωτοβουλία, να υπάρξει μία ακρόαση, να γίνει δηλαδή μία συζήτηση για τις ε, συνέπειες του Brexit στον τουρισμό. Θα ήθελα να καλωσορίσω καταρχάς τα συνδικάτα που δέχθηκαν να συμμετέχουν, καθώς επίσης και όλους τους εταίρους που είναι παρόντες εδώ όπως πάντα, θα κάνω μία μικρή σύνοψη των όσων κάναμε από την προηγούμενη συνεδρίαση της Task Force και ε, τα όσα συνέβασαν εδώ στην Επιτροπή μας και μετά θα περάσουμε στο θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Μαζί με την Πρόεδρο συστήθηκε αυτή η Task Force όπως ακούσατε και στην αρχή, η πρόεδρος ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα, αλλά ούτως ή άλλως ε, είχαμε συμφωνήσει να γίνει αυτή η συνεδρίαση. Τι συνέβη λοιπόν τις τελευταίες εβδομάδες. Στις 27 Φεβρουαρίου έγινε η τελευταία συνεδρίαση της Task Force. Είχαμε έναν προσκεκλημένο τότε, ο οποίος ε, μας επενδιαφέροντα πράγματα και την επόμενη μέρα ο πρόεδρος Ταγιάννη στις 28 του μηνός υπέγραψε τη Συμφωνία Συνεργασίας, ε, κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν και το οποίο ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Θα μπορέσουμε βεβαίω να το συζητήσουμε και στο μέλλον το θέμα αυτό και ελπίζουμε να μπορέσει να συνεχιστεί η συνεργασία και στο μέλλον και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι της Επιτροπής ε, θα δείξουν ενδιαφέρον. Συνεδρίασε και το VTTC την προηγούμενη εβδομάδα στο Buenos Aires. Εκεί εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, και, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί δεν υπήρχε άλλος εκπρόσωπος και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι υπήρχαν ναι, μία σειρά από οργανώσεις παρούσες, είχαμε και διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες ε, παρουσίασαν μία σειρά από πολύ σημαντικές ε, πρωτοβουλίες, ε, κυρίως όσον αφορά τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Και εδώ θα πρέπει να ε, ασχοληθεί με το θέμα αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητήθηκε επίσης και το θέμα της ασφάλειας των ταξιδίων. Έγιναν κάποιες πρωτοβουλίες από αυτό και υπήρχε και ένα δελτίο τύπου σχετικό του VTTC. Έγινε στη Βουλγαρία και Συμβούλιο ε, Τουρισμού πριν από μερικές εβδομάδες στα πλαίσια της Βουλγαρικής Προεδρίας και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά συγχαίρω τη Βουλγαρική Προεδρία διότι διοργάνωσε πραγματικά μια εκδήλωση για τον τουρισμό ε, πολύ ε, καλού επίπεδου και αυτό σπανίως το είχαμε δει στο παρελθόν ελπίζω να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα το οποίο θα ακολουθήσουν ε, στη συνέχεια και οι επόμενες προεδρίες. Πραγματικά επρόκειτο για μια εξαιρετική εκδήλωση. Αυτή την εβδομάδα έχουμε συνάντηση της οργάνωσης ε, που περιλαμβάνει ε, ξενοδοχεία και εστιατόρια και θα γίνει μια συνάντηση υψηλού επίπεδου στη Βιέννα, στη Βιέννη, συγγνώμη. Και επίσης ε, να σας πω και κάτι ακόμα. Προσφάτως ξεκίνησε η λειτουργία της σελίδα European Capitals of Smart Tourism. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από πρωτοβουλία της Επιτροπής μας και επομένω θα ήθελα να επενθυμίσω και στα συνδικάτα και στους συναδέλφους ότι αξίζει τον κόπο να ε, διαδώσετε το μήνυμα και στις χώρες σας διότι έτσι θα μπορούμε να αποφασίσουμε και θα μπορέσουμε να δώσουμε και τα πρώτα βραβεία για αυτές τις ε, έξυπνες ε, τουριστικές πρωτεύουσες. Έγινε και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Κοινοβούλιο και θα υπάρξουν φυσικά και άλλες εκδηλώσεις ε, και είμαι βέβαιος ότι θα σας πούν και οι συνάδελφοι και ο Εντουάρντ θα ε, ενημερώσει σχετικά. Τώρα, το Φεβρουάριο το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα στο οποίο ζητούμε ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού για τον τουρισμό έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχουν ε, γίνει τα πρώτα στάδια, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κερδίσει, γιατί ακόμα το τουριστικό λόμπι, δεν έχει τόσο μεγάλη ισχύ στις, ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και νομίζω ότι και ο κλάδος και το κοινοβούλιο κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δυστυχώς ε, είναι ελάχιστες οι απαντήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι από την Επίτροπο Μπιανκόφσκα που είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά στον προπολογισμό, μαζί με την κυρία Τσαπαρντέλ, την κυρία Ντεμόντε και άλλους συναδέλφους έχουμε ξεκινήσει ε, και στείλαμε μια επιστολή στον Πρόεδρο Γιούνκερ και στον Επίτροπο Έτιγκερ ε, και ζητούμε ο τουρισμός να συμπεριληφθεί καταλήλως στον προπολογισμό. Ξέρω εδώ ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου προσπαθούν να πιέσουν και αυτοί με τη σειρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ λοιπόν να συνεχίσετε τη βοήθειά σα. Και τώρα κάτι ακόμα όσον αφορά τι θεωρήσει διαβατηρίων. Ε, ξεκίνησε ένα νέο γύρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα πολιτική για τι θεωρήσει διαβατηρίων και το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη διευκόλυνση που σκοπεύουν να παρέχουν και θέλουμε να έχουμε και μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή ε, Τραν αλλά πρέπει να πω ότι δυστυχώς ε, αρκετές από τις προτάσεις μας ε, δεν συμπεριλήφθησαν. Υπάρχουν όμως μια σειρά από πρωτοβουλίες που είχαμε προτείνει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελήφθησαν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε λοιπόν αυτά να περιλαμβάνονται στον νέο κανονισμό για τις θεωρίες διαβατηρίων. Παραδείγματο χάρη ε, θεώρηση πολλαπλών εισόδων και φυσικά όποιος έχει κάτι να μας πει επί του θέματος μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Περνάμε τώρα στο θέμα της σημερινής ακρόασης. Να ευχαριστήσω την, πρόοδο, την Πρόεδρο που δέχτηκε αυτή την ε, πρόταση, να μπορέσουμε δηλαδή να συζητήσουμε για τις συνέπειες του Brexit στον τουρισμό, διότι είναι κάτι το οποίο δεν συζητιέται πάρα πολύ στις μεγάλες πολιτικές συζητήσεις. Ε, έχουν υπάρξει διάφορες ε, τρικυμίες για τις σχέσεις μεταξύ Λονδίνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ελάχιστα έχει πει κανείς για τον τουρισμό. Και ε, δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι δεν υπάρχει αντίκτυπος για τον τουρισμό. Ίσα ίσα είναι πολύ σημαντικός ο αντίκτυπος, διότι... Ε, ε, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, που πρέπει ήδη να έχουν προγραμματίσει κάποια πράγματα ε, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν πρέπει να γνωρίζουν πώς θα πρέπει να οργανώσουν κάποια πράγματα για την περίοδο μετά το Brexit. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αποφασίσαμε σήμερα να μιλήσουμε με κάποιους ειδικούς. Να σας πω κάποια στοιχεία. Το 76% των Βρετανών, περίπου 47 εκατομμύρια άνθρωποι, επιλέγουν ευρωπαϊκούς προορισμούς κατά κύριο λόγο. Και περίπου το 50% ε, αυτών που φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αποχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για πολύ μεγάλο μεγάλο αριθμό ατόμων. Επομένως δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό τον ε, τομέα στην ασάφεια. Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στου ε, προσκεκλημένου μα. Έχουμε διάφορου εμπειρογνώμονε. Ο πρώτο θα είναι ο κύριο Τόμα Τζένκινς, ε, ο οποίο είναι εκτελεστικός ε, διευθυντής ε, του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρισμού. Θα ήθελα να ζητήσω να περιοριστείτε στα 7 λεπτά, εάν έχω υπολογίσει σωστά το χρόνο, και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Τόμας, παρακαλώ. Thank you. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα να έχω τη δυνατότητα να σας μιλήσω. Λέγομαι Tom Jenkins ε, και είμαι εκτελεστικός διευθυντής του, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Τουρισμού. Πολλές, ε, πολύ σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί της Ευρώπης ε, βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και φυσικά μας απασχολεί πολύ το Brexit. Το Brexit μου θύμισε τα λόγια του Τσέρτσιλ. Όλα τα πράγματα στην Ευρώπη ξεκινάνε με λόγια του Τσέρτσιλ. Ε, περιέγραψε την κατάσταση στη Ρωσία ως ε, ένα ένιγμα τυλιγμένο σε μυστήριο που βρίσκεται μέσα σε ένα βαγρύφο και η απάντηση ποια ήταν ε, ε, τα ρωσικά ίδια συμφέροντα. Βέβαια στο Brexit είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς εθνικά συμφέροντα. Ε, το ανέκδοτο που λένε στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή λέει ότι σε σχέση με τις προτάσει που δεν μπορεί να αρνηθεί κανεί, λένε ότι το Brexit είναι μια πρόταση που δεν μπορεί να καταλάβει ο ε, αποδέκτης. Ε, και το Brexit μοιάζει με χήμερα. Η χήμερα δύο πράγματα είναι. Είναι ένα υβρίδιο ε, ανάμεσα σε λιοντάρι φίδι και ε, ε μια γίδα που ε, βγάζει φλόγες, ε, σημαίνει όμως και φαντασίωση και αυτό ακριβώς είναι το Brexit αυτή τη στιγμή. Δεν έχει την ε, νοητική βάση που συνδέεται με τα γεγονότα. Ως επιχειρήσεις όμως αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα στην, ε, στον τουρισμό. Στην παρουσίαση αυτή μου ζητάτε να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε όμως τίποτα ουσιαστικό στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Η μεγαλύτερη προσθήκη αξίας στον τουρισμό είναι οι πωλήσει. Ε, έτσι δίνει αξία 15 ε, ε, με 20 λίρες σε ένα κομμάτι χαρτί. Το ίδιο με, στην κράτηση δωματίου ξενοδοχείου που του δίνει αξία 200 με 300 λίρες. η ανικανότητα του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρώπη θα είναι καταστροφικό για τις επιχειρήσεις. Δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο στον τουρισμό είναι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν και με σκληρό Brexit θα έχουμε καταστροφικό αντίκτυπο και για τους ανθρώπους για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουριστικό τομέα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε, στο 70, ε, υπάρχουν επιχειρήσεις ε, τουριστικές στο Ηνωμένο Βασίλειο που το 70 με 80% των ανθρώπων που εξυπηρετούν τους πελάτες είναι υπήκοοι άλλων χωρών και όχι του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Brexit λοιπόν θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και αυτό δεν είναι καλό για τις επιχειρήσεις. Ήδη βλέπουμε σημαντική μείωση στην ε, ποικιλία και τον όγκο των ε, αιτήσεων και βλέπουμε επίσης ε, περιορισμό στις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι θα γίνει με την αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου με το Brexit. Υπάρχει τεράστιο αδιέξοδο όσον αφορά την εναρμόνιση στον τομέα αυτόν. Όπως και άλλοι τομείς ε, δεν θέλουν ξεχωριστούς κανόνες. Κανείς δεν θέλει δύο ξεχωριστές σειρέ κανόνων. Εάν λοιπόν δούμε κατακαιρματισμό αντί για εναρμόνιση, μπορούμε να περιμένουμε τις επιχειρήσεις να δημιουργούν παρακλάδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι τέσσερι ελευθερίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τι τουριστικέ επιχειρήσει. Ε, θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν το προσωπικό του εκεί που υπάρχει ζήτηση. Και κάποιοι βλέπουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, μια δύναμη μεταρρύθμισης που δημιουργεί όλο και καλύτερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις. Έχουμε την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια που θα τεθεί σε ισχύ σε δύο μήνες από τώρα είναι ήδη παροχημένη. Διότι προσπαθεί να μεταρρυθμίσει τον τομέα των ταξιδίων και την κατανομή τους, αλλά αυτό έχει αλλάξει δραματικά στο διάστημα εκπόνησης της οδηγίας αυτής και πρέπει να ξεκινήσουν τώρα οι συζητήσεις για την διαμόρφωση της τρίτης δέσμης μέτρων, για ε, της τρίτης οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια και το Ηνωμένο Βασίλειο πώς θα συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Θα επηρεάσει την ανάπτυξη του Brexit. Ναι, πολύ απλή απάντηση. Εμείς προσπαθούμε να πουλήσουμε το εισαγωγικών την ε, Ευρώπη. Είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο πακέτο που έχουμε είναι ε, ταξίδι Λονδίνο-Παρίσι. Οτιδήποτε αυξάνει το διοικητικό άχθος θα μειώσει την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ποιο λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα προς τους διαπραγματευτές όπως όλοι οι άνθρωποι, όπως όλοι οι επιχειρηματίες, θέλουμε διατήρηση του status quo για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα. Και ε, ελπίζουμε να δούμε εκ Θεό. Τι μορφή θα έχει αυτός ο ε, ε, εκ Θεό. Μπορεί να έχει τη μορφή ακριβώς ε, του ε, εθνικιστικού εγωισμού, των εθνικών συμφερόντων. Ευχαριστώ. So much, uh, Tom. Σε ευχαριστούμε, Τόμ. Τέλεια. Και ακριβώς μέσα στο 7 λεπτό. Περνάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Μαρκ Τάντσερ εκτελεστικός διευθυντής ε, της ε, Ταξιδιωτικής Ένωσης ε, ΑΠΤΑ, Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Γραφείων Προσφερών των Πακέτων Διακοπών. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για όσους δεν γνωρίζουν την ΑΠΤΑ, είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική ένωση. Έχουμε 1.200 μέρη και 40 δις τζίρο εργασιών. Και μάλιστα έχουμε ταξίδια από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, ε, κυρίως όμως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σημαντικό δημόσιο προφίλ και εμπορικό και όταν αναγκέρθηκε το δημοψήφισμα πήραμε τις αποστάσεις και δεν δώσαμε οδηγίες, αλλά ε, θα είναι μεγάλος ο αντίκτυπος του Brexit και για τις επιχειρήσεις της ταξιδιωτικές και για τους τουρίστες. Ε, και μας μας αρέσει το status και ή μέχρι τώρα ρυθμίσει επέτρεψε στην άνθηση του τουρισμού και για τα μέλη μας, του ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλλά και για τους προορισμούς. Και τα μέλη μας τουλάχιστον δεν ε, έχουν πρόβλημα με τους κανονισμούς που διέπουν τον τουρισμό, γιατί δημιουργούν και ενισχύουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Ε, σας είπε ο προλαλής σας στην τάξη μεγέθους ε, των ε, την οικονομική για την οποία μιλάμε. Έχουμε τη μεγαλύτερη αγορά, 53 εκατομμύρια ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, 37 δισεκατομμύρια ήταν ε, η μεικτή ε, προστιθέμενη αξία, 860.000 απασχόληση, 340.000 επιχειρήσεις που, στη, που στηρίζονται ε, στους τουρίστες και 28 δισεκατομμύρια ε, στις 7 οικονομίες ε, τις ηλιόλουστες. Οπότε τεράστιες οικονομικές δραστηριότητες, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τις χώρες ε, προορισμού, προς τις οποίες δηλαδή μεταβαίνουν, ταξιδεύουν οι, οι ε, ταξιδιώτες, οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια είναι τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας και θέλαμε να διαφυλάξουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Καταρχήν, ε, η πολιτική αεροπορία. Φυσικά, κυρίως με αεροπορικά έρχονται οι τουρίστες και φεύγουν οι τουρίστες μας από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τους προορισμούς. Οπότε ε, με τη μείωση του κόστους ε, άνοιξαν και νέοι προορισμοί που στο παρελθόν ήταν απρόσιτοι. Θα θέλαμε και αυτή την κατάσταση να τη διατηρήσουμε και να την προωθήσουμε προς το αμοιβαίο όφελος ε, της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, έχουμε διακίνηση βασικών εργαζομένων, στηρίζοντας τους επιχειρηματίες, τους ε, ταξιδιωτικούς πράκτορες, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Θέλουμε και αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα να τα διατηρήσουμε και να κρατήσουμε αυτή την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων που ήταν πολύ σημαντικό ε, και πολύ σημαντικό και για μας ε, την τουριστική βιομηχανία. Τώρα, ελεύθερη ροή από τα σύνορα χρησιμοποιούμε την ίδια διανομή με ε, τις ίδιες υποδομές με τη, το, τη διακίνηση εμπορευμάτων. Οπότε, αν δεν έχουμε τελωνιακή ένωση, θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου στις διαπραγματεύσεις, τον αντίκτυπο που θα έχει το Brexit στον τουρισμό, αν έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στα σύνορα με ελέγχους. Επίσης, θέλουμε να διαφυλάξουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όπως με κανονισμούς για τα πακέτα οργανωμένων ταξιδιών, αλλά με την ε, ηλεκτρονική κάρτα ε, ασφάλειας υγείας. Υπάρχει αμοιβαιότητα με την αντίστοιχη Βρετανική κάρτα. Επίσης και εμείς στηρίξετε με την κατάργηση των, τελών περιαγωγής. Ήταν πολύ θετικές όλες αυτές οι εξέλιξεις. Όλα αυτά είναι σημαντικά και κέρια για τη διατήρηση του τουρισμού και της άνθησης του τουρισμού. Τώρα, αυτά είναι όσα θέλουμε να διατηρήσουμε. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι ένα σκληρό Brexit. Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο χωρί συμφωνία για την αεροπορία, αυτό θα ήταν αδιανόητο για μα. Καταστροφικό σενάριο. Κάτι άλλο που θέλουμε να αποφύγουμε είναι μία ρήξη και μία βεβαιότητα ώστε ούτε οι τουρίστες ούτε οι επιχειρηματίες να μην γνωρίζουν ποια θα είναι η κατάσταση από το χρόνο και μετά. Ποια είναι η στρατηγική μας για να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας και τις προτεραιότητες μας. Θα κάνω μια ανάλυση, να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να συνειδητοποιήσει και η κυβέρνηση τη σημασία την οικονομική και κοινωνική σημασία ε, που θα έχει το Brexit και έχουμε και διμερείς επαφές με τις ε, ε, περισσότερο πληγέντες προορισμούς. Και έχουμε συμφωνήσει σχεδόν απόλυτα ότι ο τουρισμός είναι πολύ θετικός οικονομικά, και θα πρέπει να τον διατηρήσουμε. Φυσικά ε, τα οικονομικά επιχειρήματα και τα επιχειρηματικά πολλές φορές απάδουν από τα πολιτικά. Και μέχρι στιγμής η κυβέρνηση ήταν πολύ πιο θεωρητική παρά συγκεκριμένη ως προς το μέλλον αυτών των ρυθμίσεων. Πάντως η Πρωθυπουργό άρχισε να περιγράφει κάποιες κόκκινες γραμμές, που όμως δεν είναι και πολύ αδιάλακτες, γιατί αναφέρθηκε και ο οργανισμός για την πολιτική αεροπορία που θα πρέπει να το κρατήσουμε ε, και επίση η δικαιοδοσία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Αυτό είναι μια αναγνώριση ότι δεν μπορούμε να αποκοπούμε από τέτοιες ρυθμίσεις. Ε, θα περάσουμε τώρα στη δεύτερη φάση που θα είναι κρίσιμη το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να πει επιτέλους ξεκάθαρα και να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να τα έχει όλα. Δεν μπορεί να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο, δηλαδή πλήρη πρόσβαση αλλά χωρίς κανόνες. Θα πρέπει να δούμε που θέλουμε να ενταχθούμε σε αυτό το φάσμα. Και ε, θέλουμε να είμαστε εταίροι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε διαπραγματεύσει και με το Βρετανικό κοινό. Και θα πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες η ελπίδα μου και η ευχή μου είναι ότι σίγουρα ε, θα και οι δύο πλευρές και θα κερδίσουν και θα χάσουν. Και βλέπετε πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός και για τις δύο πλευρές, γι' αυτό ελπίζω τουλάχιστον τα ωφέλη του να τα διαφυλάξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μάρκ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Γκοστάβο Μαρτινιέ από την Ισπανία, από την Βαλένθια εξ ονόματος ε, της Next Tour. Νομίζω ότι όλοι εδώ στην αίθουσα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την Next Tour και γι' αυτό ακριβώς ε, σας προσκαλέσαμε κιόλας ε, για να ακούσουμε την άποψή σας. Παρακαλώ, Γουστάβο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω την παρουσίασή μου στα ισπανικά δεν ξέρω αν θα είμαι τόσο ακριβής όσο οι προλαλήσαντες και θα τηρήσω τα 7 λεπτά, αλλά θα προσπαθήσω. Η ιδέα είναι να προσθέσουμε και εμείς το λιθαράκι μας στη συζήτηση και να σας παρουσιάσω και την ε, ε, περιφερειακή άποψη. Εγώ εργάζομαι για την ε, αυτόνομη περιοχή της Βαλένθια ε, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ισπανίας και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε λίγο την περιφερειακή άποψη. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τον Brexit, είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τον Brexit, αλλά αυτό το οποίο θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε ευθύ εξ αρχή είναι ότι πολλά από τα σημεία τα οποία αποσχολούν τις διάφορες περιφέρειες περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων να σας πω ότι καταρχήν πολλές ε, περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θεώρησαν θετική αυτή την πρώτη προκαταρκτική συμφωνία. Ε, σίγουρα βέβαια κρεμούν πάρα πολλά και πολύ δύσκολα. Πρέπει να δοθεί ε, νομική οντότητα στο θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών, το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η αναγνώριση των προσόντων. Κάποια από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί. Και όπως πολύ σωστά λέει η έκθεση που καταρτίστηκε από κοινού, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα από πλευράς ε, περιφερειών ε, και στην Επιτροπή των Περιφερειών πιο συγκεκριμένα, πολλές εθνικές αντιπροσωπείες ε, ασχολήθηκαν με έγγραφα και είπαν τι τους ανησυχεί όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit. Έγιναν πολλές συζητήσεις δημοσιεύτηκαν και αναλύσεις και η τελευταία καινοτομία είναι η σύσταση μιας ε, διαπεριφερειακής ομάδας για τον Brexit. Έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές, ε, έχει 20 περιφέρειες που συμμετέχουν και ο στόχος είναι να διευκολύνουν το διάλογο. Το διάλογο διότι όλοι γνωρίζουν ότι το Brexit θα έχει έναν περισσότερο ή λιγότερο αρνητικό αντίκτυπο, δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα τα πράγματα θα αλλάξουν. Η ιδέα λοιπόν αυτής της διοργανικής ομάδας είναι να προσπαθήσουμε προσπαθήσουν να ε, απορροφήσουν όσο δυνατόν περισσότερο τους κραδασμούς της, ε, ε, των συνεπειών σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, επίσης, πέραν αυτών, υπάρχουν και διαπεριφερειακά δίκτυα τα οποία δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες και αυτές ασχολούνται με τον αντίκτυπο του Brexit. Μεταξύ αυτών, αναφέρουμε το ERIN, για παράδειγμα, που είναι ένα δίκτυο το οποίο ασχολείται με την καινοτομία και την έρευνα ή το CRPM που είναι η διάσκεψη των ε, περιφερειακών και θαλάσσιων περιοχών που και αυτοί ε, με τα μέλη της περιφέρειας που συμμετέχουν κοιτάνε να δούνε πώς ε, θα διαμορφωθεί ο αντίκτυπος. Ξεχνάω και την παρουσίασή μου, βλέπετε. Είμαστε στη διαφάνεια 4. Και ζητώ συγγνώμη. Στην περίπτωση των δικτύων, λοιπόν, υπάρχει η μελέτη ε, της NextEar και της ERPM. Η NextEar ασχολείται περισσότερο με τον τουρισμό. Είναι ένα δίκτυο που ασχολείται για, με τον ανταγωνιστικό και βιώσιμο τουρισμό. 37 περιφερειακές αρχές, 33 συνδεδεμένες ε, περιφέρειες και από τις περιφερειακές αρχές που διαχειρίζονται τους προορισμούς, ε, ε, αλλά έχουμε επίσης και συμμετοχή του πανεπιστημιακού τομέα και του τομέα της έρευνας. Έχουμε πάνω από 10 χρόνια δραστηριότητα, το γνωρίζετε ίσως αυτό, και προέκυψε ακριβώς από την ανάγκη που είχαν οι περιφέρειες να συνεργαστούν για να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Εδώ σήμερα έχουμε αρκετά μέλη της Next Tour, πολλά εξ αυτών ε, τρία πιο συγκεκριμένα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και έχουμε και τη Σκοτία. Και η Σκοτία έχει παρουσία εδώ σήμερα. Και τώρα, δύο λόγια παραπάνω για την Ex ε, Tour. Από πλευράς Ισπανικών περιφερειών, εμείς συντονίζουμε και την Ισπανική Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών. Οι Ισπανικές Περιφέρειες έχουν εκπονήσει ένα έγγραφο κοινή θέση ε, και λένε ποιες είναι οι συνέπειες που μπορούμε να προκύψουν από το Brexit. Όπως και στον τομέα των υπηρεσιών, για να διακρίνω κάποια από αυτών, ε, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία θα είναι ε, λόγω της απώλειας δικαιωμάτων. Πράγματα τα οποία ήδη ε, μας απασχόλησαν στην πρώτη διαδικασία της συμφωνίας. Ε, θα υπάρχουν ευρωπαϊκές και βρετανικές επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα, το θέμα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ε, ψηφιακές υπηρεσίες, το ανέφερε προηγουμένως το θέμα του roaming ο προλαλής ε, και ε, αρκετά άλλα. Στις ισπανικές περιφέρειες της απασχολεί επίσης σχετίζεται και με τον τουρισμό, το θέμα των εμπορικών ανταλλαγών. Υπάρχει ένα αρνητικό πανόραμα που προβλέπει την πιθανή ε, ρίκνωση της ε, Βρετανικής οικονομίας ε, και δημιουργούν μια πολύ ανησυχητική εικόνα φυσικά. Ε, επίσης ε, πλήττεται και ο τομέας των ακινήτων, η αγορά κατοικιών στην Ισπανία έχει ήδη πληγεί και δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά μεν πώς θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, αν θα είναι σκληρό ή πιο ήπιο το Brexit, αλλά αυτό σίγουρα που γνωρίζουμε είναι ότι τη στιγμή που γινόταν η ψηφοφορία είναι ότι υπάρχει ήδη κάποιος αντίκτυπος, για παράδειγμα στον τομέα των ακινήτων. Οι αγοραπολισίες ε, ε, και αυτό είναι παράδειγμα που σας δίνω για την περιφέρεια τη, ε, της Βαλένθια, ήδη υπάρχουν συνέπειες ε, και νιώθουμε το Brexit ήδη στον τομέα των αγοραπολασιών ακινήτων. Και αυτό είναι σημαντικό διότι πολλές κατοικίες αγοράζονται από Βρετανούς ε, πολίτες και το έχουν ως δεύτερη κατοικία και αυτό εμείς το αποκαλούμε τουρισμό κατοικίας δηλαδή ζουν ένα διάστημα το χρόνο εκεί και θεωρούνται εξοχικές κατοικίες αυτές. Ε, υπάρχουν πολλοί Βρετανοί, κυρίω στην περιοχή της Βαλένθια και πρέπει να σα πω ότι είναι αρνητικό το οικονομικό πανόραμα και σίγουρα αυτό ε, θα πλήξει και την αγοραστική τους δύναμη και φυσικά αυτό θα έχει συνέπειες. Όσον αφορά τον τουρισμό, θα υπερβώ βέβαια τα 7 λεπτά, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πρώτη αγορά ε, τουριστών ε, προς την Ισπανία. Αν υπάρξει κάτι αρνητικό, σημαίνει ότι θα επιλέγουν διαφορετικούς προορισμούς, εναλλακτικούς προορισμούς εκτός Ευρωζώνης. Το ίδιο θα συμβεί αν αυτή η διαπραγμάτευση τελικά έχει και νέους διοικητικούς ελέγχους. Οποιοδήποτε επιπλέον έλεγχος για να εισέλθει στην Ισπανία ένας Βρετανό πολίτη, σημαίνει ότι θα υπάρχει επιπλέον κόστος. Και φυσικά αυτό που θα ε, αλλάξει σίγουρα είναι ότι θα αλλάξει η δυναμική μεταξύ των ε, αεροπορικών επιχειρήσεων εταιριών low cost ε, και όλες τις τουριστικές δραστηριότητες οι οποίες ε, προσφέρουν στην αλυσίδα αξία του τουρισμού, διότι δεν έχουμε απλώς κάτι συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο θα κλιμακωθεί σε γενικό επίπεδο. Όσον αφορά τη Βαλένθια, και εδώ έχουμε και την επόμενη διαφάνεια, και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως σας είπα, είναι ο κύριος ε, ε, Αριθμό τουριστών που έχουμε και εδώ βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά των ακινήτων. Έχει υπάρξει επιβράδυνση από τον Οκτώβριο και αν κάνουμε σύγκριση σε επίπεδα τριμήνου, το πρώτο τρίμηνο του 2016 με το πρώτο τρίμηνο του 2017 που έχουμε τα στοιχεία, το αποτέλεσμα είναι αρκετά ανησυχητικό, διότι έχουμε μια πτώση της τάξης του 31% για αυτό το τελευταίο τρίμηνο. Ε, το θέμα της υγείας ε, για τους ε, Βρετανούς που περνούν μεγάλο διάστημα στην Ισπανία είναι επίσης σημαντικό. Και επίσης μας ενδιαφέρει και πώς μπορεί να επηρεάσει τον κλάδο η μείωση της συχνότητας των αεροπορικών πτήσεων. Αν για παράδειγμα μειωθεί η συχνότητα, στο αεροδρόμιο του Κάντε έχουμε 13 εκατομμύρια ετησίως τουριστών, από τα οποία τα 6 εκατομμύρια είναι Βρετανοί σύγκριση μεταξύ του 2016 και 2017 ε, και σε επίπεδο του κάθε μήνα μας δείχνει ότι υπάρχει μείωση. Υπάρχουν κάποια περαιτέρω παραδείγματα σε επόμενες διαφάνειες, ε, η περίπτωση της Ανδαλουσίας για παράδειγμα, που μας έδωσε και αυτή τις πληροφορίες της. Η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας θεωρεί ότι μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι κατά 1% αρνητική η συνέπεια για το ΑΕΠ. Και αυτό ε, σημαίνει ότι οι συνέπειες του Brexit θα ε, επεκταθούν για τουλάχιστον 10 χρόνια. Επίσης, ε, θα πρέπει να πω για την περίπτωση της Ανδαλουσίας ότι υπάρχει και το θέμα του Κυβραλτάρ, που την χάνει διαφορετικές μεταχείρισεις εντός των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε επίσης και τη συμβολή της περιοχής της Φλάνδρας, που έχει σημαντική ροή τουριστών από τη Βρετανία και ήδη αντιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ότι ε, σήμερα οι τουριστικές ροές έχουν μειωθεί κατά 1,4% και αναμένουν να πέσει μέχρι και το 10%. Ε, και επίσης έχουμε κάποιες συστάσεις τις οποίες θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε. Το πρώτο είναι να μην υπάρχει σκληρό Brexit ή ήπιο Brexit, αλλά ένα Brexit το οποίο θα είναι φιλικό προς τους πολίτες. Ε, διότι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα νιώσουν τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το Brexit θα πρέπει να είναι ένα ε, Brexit φιλικό προς τους πολίτες. Ε, Επίση, να συμμετέχει και η Επιτροπή των Περιφερειών και οι περιφερειακές κυβερνήσει ε, στις διαπραγματεύσεις μέσω των εθνικών κυβερνήσεων, διότι πολλές από αυτές τις διαπραγματεύσεις έχουν να κάνουν με αποκλειστικέ του αρμοδιότητε. Οι περιφερειακέ αρμοδιότητε είναι πολύ σημαντικέ και οι περιφέρειε απουσιάζουν. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για να μετριάσουμε τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες. Αυτό και για την επόμενη ε, τη δημοσιονομική περίοδο και θα πρέπει σίγουρα να συμπεριλάβουμε εδώ και το θέμα του πώς ε, μπορούμε να έχουμε τις πιθανές συνέπειες και πώς μπορούμε να μετριάσουμε αυτές τις συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, υπάρχει το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης και της αναγνώρισης ε, των μισθών και συντάξεων και επίσης να σκεφτούμε οποιοδήποτε εμπόδιο, είτε είναι ε, ε, φορολογικό, μη φορολογικό, διοικητικό, ε, γραφειοκρατικό που δεν επιτρέπει τις εμπορικές σχέσεις, θα πρέπει να το εξετάσουμε και να διορθωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε τώρα από την Βαλένθια στην Σκοτία. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάκομ Ράφρεντ ε, από την Visit Scotland. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Uh, Λέγομαι Μάκομ Ράφρεντ, είμαι εκπαιδευτικός διευθυντής της Visit Scotland και είμαστε ε, ο Εθνικός Φορέας Τουρισμού της Σκοτίας. Στην εντολή μας περιλαμβάνονται εκδηλώσεις, ο αθλητισμός, ε, πολιτισμός, ο ε, τουρισμός ε, των επιχειρήσεων και άλλα. Και ο τουρισμός ως ε, στοιχείο κλειδί της τουριστικής οικονομίας φαίνεται από το ότι είναι ένας από τους τομείς ανάπτυξης στην Σκοτία. Ε, από το 2008 μέχρι το 2014 ο τουρισμός αναπτύχθηκε κατά 42% στη Σκοτία, ενώ η απασχόληση το 2015 αυξήθηκε κατά 11%, δηλαδή αντιπροσωπεύει το 9% ε, του, της συνολικής απασχόλησης και αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό από τότε που ξεκίνησαν ε, οι σχετικές ε, στατιστικές. 14,3 ε, επισκέπτες ε, διανυκτερεύσεις ε, είχαμε και 142 εκατομμύρια μονοήμερες εκδρομές, συνολικά 4,9 εκατομμύρια λίρες. Με τον αντίκτυπο στην εφοδιαστική αλυσίδα ε, συνολικά ο τουρισμός αντιπροσωπεύει 11 δισεκατομμύρια λίρες ε, στην Σκοτία. Ε, Εξαρτόμαστε λοιπόν απολύτως από την υγεία του τουριστικού τομέα περισσότερο από άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και με το Brexit θα έχουμε καταστροφικές συνέπειες στον τουρισμό της Σκοτίας. Οι τουρίστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Για μας το 54% των ε, τουριστών προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία αποτελούν τον ε, μέσο όρο για τρία χρόνια, 2014 έως 2016. Αυτό σημαίνει 1,4 ε, εκατομμύρια ταξίδια το χρόνο από πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δαπανούν περίπου 710 εκατομμύρια λίρες ε, στη Σκωτία. Πάνω από το μισό προέρχονται από Γαλλία, Γερμανία και τις κάτω χώρες ε, και βλέπουμε μάλιστα επανειλημμένες επιστροφές στην Σκωτία. Ε, μεγάλη το μεγαλύτερο τμήμα είναι ηλικίες 35 έως 45 ετών, αλλά είδαμε και μεγάλη αύξηση ε, στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία 45 έως 54 ετών. Θέλουμε να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές, να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές με συναδέλφου ε, στη Ρωσία σε τομείς όπω είναι ο κοινωνικό τουρισμό, ε, ο προσβάσιμος τουρισμός, η οργάνωση εκδηλώσεων και γενικά στο ΜΑΚ marketing. Και όσον αφορά τις εταιρικέ ε, σχέσεις, ε, συμμετέχουμε ε, στον οργανισμό DNA. Αυτό σίγουρα δεν πρόκειται να αλλάξει στο μέλλον. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχαμε στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις με εταίρους στην Ευρώπη που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε στη συνέχεια άσχετα από το τι θα γίνει. Η ίδια η απόφαση του Brexit ε, θέτει σημαντικά ερωτήματα για το μέλλον ε, της οικονομίας αλλά και του τομέα φιλοξενίας και του τουρισμού ιδιαίτερα. Πολλά παραδείγματα ανέφεραν οι τρεις προηγούμενοι ομιλητές, ε, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν. Αλλά σε σχετική έρευνα φάνηκε ότι το 75% των επιχειρήσεων θα ε, είχαν αύξηση του κόστους ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ε, και οι επιχειρήσεις περιμένουν ότι αυτό ε, έχει να κάνει με την ισοτιμία της ΛΥΡΑΣ, αλλά και λόγω της αλλαγής του καθεστώτος υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βρετανία. Επίσης υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και σε άλλους τομείς και ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Μετά το δημοψήφισμα για ε, το Brexit το 2016 είδαμε αρχική ε, πτώση της λίρας ε, κάτι που οδήγησε σε αύξηση της αύξησης, αλλά το βραχυπρόθεσμο κέρδος ε, δεν ε, προβλέπει απαραίτητα το μέλλον. Όσον αφορά λοιπόν την ε, φήμη της Σκοτίας μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, δεν βλέπουμε να υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος. Αυτό αντικατοπτρίζει και όλη την δουλειά που έχει γίνει εντός της Ευρώπης ε, για, την, για να διαβεβαιώσουμε τους ε, τουρίστες ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά σε αυτό. Οποιαδήποτε πρόσθετα εμπόδια, ε, υψηλότερο κόστος ε, ή θεωρήσεις για παράδειγμα θα πρέπει να αποφευθούν και έτσι φτάνουμε στην ε, ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού το οποίο αναφέρθηκε. Ε, αυτή είναι σίγουρα η μεγαλύτερη ανησυχία για τον ε, τομέα φιλοξενίας και τουρισμού στην Σκοτία. Και οι προβλέψεις είναι δυσμενείς. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν επαρκή επαρκές ε, εργατικό δυναμικό. Πάνω από 56.000 άνθρωποι απασχολούνται στον, ε, στα ξενοδοχεία και σχεδόν 124.000 αν συμπεριλάβουμε και τα εστιατόρια και σχεδόν 65.000 στον ε, τομέα τροφοδοσίας, στο catering. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ε, ποσοστό ε, υπηκών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, και άλλωστε το 4,1% του πληθυσμού της Σκωτίας είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 290.000 συνολικά. Ε, απασχολούμε ανθρώπους από πολλές διαφορετικές χώρες ε, και όλοι αυτοί συμβάλλουν με τις ειδικές τους αξιότητες ε, στην ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι σαφές ότι η πιθανή απώλεια των εργαζομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αντίκτυπος και οι διάφορες ομάδες συμφερόντων πιέζουν την κυβέρνηση ώστε να ληφθούν επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα του τομέα του τουρισμού στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνοψίζοντας λοιπόν, όποιος και αν είναι ο αντίκτυπος του Brexit, η Visit Scotland θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους ε, εταίρους μας ε, για να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε τους φίλους μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ανταποκριθούμε με θετικό πνεύμα στη, στα γεγονότα. Άλλωστε ζήσαμε και στο παρελθόν οικονομική ύφεση και ε, την ε, στάχτη από το Ισλανδικό ηφαίστειο. Ε, πάντως στο πλαίσιο του τουρισμού όλοι οι προορισμοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Αλλαγές στις ανάγκες των καταναλωτών, αλλαγές στην τεχνολογία Θέλουμε λοιπόν να φροντίσουμε όχι μόνο να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, αλλά και βιώσιμοι και η Σκοτία θα συνεχίσει να είναι πρόθυμος εταίρος για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ώστε όλοι στην Ευρώπη να μπορέσουμε να καλύψουμε τις μελλοντικές ανάγκες του τομέα μας. Σας ευχαριστώ. Thank you so Σας ευχαριστούμε. Και ελπίζω ότι και μετά το Brexit θα συνεργαστούμε γιατί η Visit Scotland είναι από τους πιο ενεργούς φορείς ε, στον ευρωπαϊκό τουρισμό, οπότε θα σας χρειαστούμε και μετά τον Brexit και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ο Νάιτζελ Μόργαν είναι ο τελευταίος μας ε, ομιλητής, είναι πρόεδρος του Τμήματος Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Σόνση. Έχετε το λόγο κύριε Μόργαν. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για την πρόσκληση σε αυτή την ακρόαση. Ε, νομίζω ότι τα πλονεκτήματα του να μιλάει κανείς τελευταίος είναι ότι διαπιστώνει τα κοινά σημεία με τους προλαλήσαντες. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Θα ήθελα πρώτα να υπογραμμίσω κάτι που είπαν και οι προλαλήσαντες, ότι Σίγουρα ο τουρισμός είναι κινητήρες μοχλός της οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης ε, και της κοινωνικής συνοχής. Και μάλιστα ο τουρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ε, είναι αλληλένδετη. Δεν χρειάζεται να επισέλθω σε λεπτομέρειες στο στατιστικό στοιχείο γιατί ήδη πολλά ακούσαμε για την έντονη αλληλεπίδραση των οικονομιών μας και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών μας. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικά βασικά στοιχεία. 8 από τους 10 8 ε, από τις 10 βασικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ευρωπαϊκές και περίπου το 50% των δαπανών γίνεται σε αυτές. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ε, πού πηγαίνουν οι Βρετανοί υπήκοοι. Ακούσαμε ήδη λεπτομέρειες για τα συνολικά νούμερα. Και νομίζω ότι είμαστε ήδη στη φάση όπου χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η Κύπρος ε, εκφράζουν ήδη ανησυχία για, τη, για τους μειωμένους αριθμούς Βρετανών τουριστών ε, που φοβούνται ότι θα σημειωθούν στο μέλλον. Και ένας από τους βασικούς λόγους για αυτό το βαθμό εξάρτησης ε, είναι η ενιαία αγορά. Επόμενη διαφάνεια. Για να υπογραμμίσω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, ε, ο τουρισμός ε, επηρεάζει ιδιαίτερα την ε, Βρετανική οικονομία και την επηρεάζει πολύ περισσότερο από ότι η γεωργία ή η αυτοκινητοβιομηχανία σε ό,τι αφορά το πολιτικό λόμπι και μία από τις προκλήσεις τις ιδιαίτερες προκλήσεις που έχουμε, κυρίως στην Ουαλία, αλλά και γενικώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι να τονίσουμε την τεράστια σημασία του τουρισμού και της οικονομίας των επισκεπτών, των ταξιδιωτών για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ε, ο τουριστικός κλάδος του Ηνωμένου Βασιλείου πάει καλά προς το παρόν. Και όπως είπε και ο Μάλκολ, είναι σημαντικό να μην στηρίξουμε το μέλλον μας σε βραχυπρόθεσμους παράγοντες. Για αυτή τη στιγμή ε, εκμεταλλευόμαστε και ευνοούμαστε από την ε, υποτίμηση της λίρας τερλίνας και την θετική για μας ε, ε, συναλλαγματική ισοτιμία. Και θα πρέπει όμως να συνεχιστεί αυτή η άνθηση του τουρισμού και να συνεχίσουν οι τουρίστες και ταξιδιώτες να υποφελούνται από τα σημερινά ωφέλη. Η επόμενη διαφάνεια είναι η αγαπημένη μου διαφάνεια σε αυτό το PowerPoint. Εγώ βλέπω το Brexit ως παγόβουνο Μερικές επιπτώσεις είναι ορατές, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότερες συνέπειες ε, του Brexit είναι αφανείς και απρόβλεπτες για πολλούς ε, ενδιαφερόμενους. Επόμενη διαφάνεια. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις του Brexit. Καταρχήν η διατήρηση του επίπεδου της σημερινής κατάστασης. Η αντιμετώπιση των πιθανών αλλαγών στις, στην αμοιβαιότητα των ρυθμίσεων για, τα ιατρικές, για τις ιατρικές δαπάνες, τα θέματα της ασφάλισης μεταξύ των κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, ε, τι θα γίνει με το τέλος αερομεταφοράς και πώς θα επηρεάσει ε, ή θα αποτρέψει τους ε, Βρετανούς ή τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, τουρίστες. Επόμενο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις ε, βασικές προκλήσεις, ε, φυσικά εγώ είμαι πανεπιστημιακός, δεν εκπροσωπώ μια οργάνωση του κλάδου, αλλά βλέπω τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις, το τοπίο είναι κάπως συγκεχημένο προς το παρόν. Ε, κάποιοι φορείς πιστεύουν ότι το Brexit ήδη έχει αρνητικό αντίκτυπο στη τουριστική φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό στηρίζεται σε έρευνες ε, ενδιαφερομένο στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Λονδίνου. Αλλά η επόμενη διαφάνεια μας δείχνει ότι στους δυνητικούς ταξιδιώτες ε, δεν επικρατεί αυτή η γνώμη. Εξαρτάται ποιο ρωτά λοιπόν κανεί ε, και σε τι στηρίζεται η έρευνα. Αν ε, ρωτήσουμε εξοκοινοτικούς επικόους, ε, αυτοί εξακολουθούν να θεωρούν ελκυστικό το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά δεν ξέρω πώς η στάση του επηρεάζεται σήμερα από την ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία της Λίρα Τερλίνα. Επόμενη ολομέλεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως σε ορισμένους τομείς. Ήδη οι Βρετανοί τουρίστες πληρώνουν περισσότερα για τις διακοπές τους στην Ευρώπη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την, ε, τις χαμηλές τιμές μεταφορές, το θέμα της, των αερομεταφορών, γιατί το πιο καταστροφικό σενάριο θα είναι να μην η συμφωνία για τις αερομεταφορές. Γιατί δεν θέλουμε να υπαναχωρήσουμε στους κανόνες του ΠΟΕ. Τι θα γίνει με τα δικαιώματα των καταναλωτών επίσης. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε τα καταναλωτικά δικαιώματα και να έχουμε ένα Brexit φιλικό προς τους πολίτες, όπως το λέμε, και να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί ως ευρύτερος ευρωπαϊκός τουριστικός προορισμός ε, και να συμπεριλαμβανόμαστε στα πακέτα ταξιδιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία θα πρέπει να τονίσουμε την πρόκληση της κινητικότητας και όσων απασχολούνται στον τομέα τουρισμού και φιλοξενίας. Σε ό,τι αφορά τους ε, Ευρωπαίους ε, υπηκόους που εργάζονται στον τουρισμό και στον τομέα της φιλοξενίας. Οριστικός αριθμός δεν υπάρχει προς το παρόν. Πάντως ο αριθμός των ε, Ευρωπαίων υπηκών ε, μεταξύ 2011 και 2016 έχει σχεδόν αυξηθεί κατά 25% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα αν δεν μπορέσουμε να εγγυηθούμε την διαμονή αυτών των ε, Ευρωπαϊκών, Ευρωπαίων επικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν διασφαλίσουμε και τις εργασιακές ρυθμίσεις που τους διέπουν. Άλλες βασικές προκλήσεις αφορούν την χρηματοδότηση. Γιατί για την Ουαλία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ε, είμαστε αποδέκτες ε, και όχι σημαντικοί κοινωνικού τμήματος των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Τι θα γίνει με τις ε, προκλήσεις του marketing, με τις προκλήσεις ανάπτυξη προϊόντων που μέχρι στιγμής χρηματοδοτούνταν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τι θα κάνουμε στο μέλλον όταν θα κλείψουν αυτέ οι χρηματοδοτήσεις. Γιατί ήδη οι τουριστικοί προπολογισμοί των, των, τοπικών κυβερνήσεων είναι κατακαιρματισμένοι και μειώνονται, οπότε οι προκλήσεις ε, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η Ουαλία είναι ε, ενδιαφέρουσα περίπτωση στη συζήτηση του Brexit, γιατί έχει βελτιωθεί η τουριστική της φήμη το τελευταίο καιρό. Αν θέλουμε όμως να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας, θα πρέπει να στραφούμε και προς τη διεθνή αγορά, που αυτή τη στιγμή είναι μόνο το 10% των επισκεπτών, αλλά 20% των δαπανών. Οπότε η Ουαλία θα έχει τεράστια πρόκληση να αντιμετωπίσει με το Brexit. Οπότε ποια είναι τα βασικά πορίσματα και τι χρειαζόμαστε από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit. Σίγουρα είμαστε κατά του σκληρού Brexit. Δεν θέλουμε ένα σκληρό Brexit, θέλουμε ένα Brexit που θα μας επιτρέψει ε, έναν τουριστικό ευρωπαϊκό κλάδο που θα ευημερεί, που θα μπορούν οι ταξιδιώτες ε, να ταξιδεύουν ελεύθερα για την αναψυχή τους και θα απολαμβάνουν τα σημερινά ε, ωφέλη και δικαιώματά τους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μόργαν. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά Φυσικά και θα ήθελα να γίνει συζήτηση και να ζητήσουμε από τους συναδέλφους ε, να λάβουν το λόγο. Η κυρία Ντεμόντε καταρχάς. Ευχαριστώ συνάδελφε, να ευχαριστήσω και τους ομιλητές για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις να ευχαριστήσουμε και τον Ίστβαν που ανέφερε τις επόμενες πρωτοβουλίες μας σε θέματα τουρισμού. Θα ήθελα καταρχάς ε, να πάω στην καρδιά του ζητήματος, ε, διότι αυτή η Επιτροπή δεν λέγεται τυχαία Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Υπάρχει στενή σχέση ε, του τουρισμού με το πώς θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Επομένως, μπορούμε να μιλήσουμε για τις αεροπορικές και το στοιχείο που έχουμε είναι ότι το 2050 θα έχουν διπλασιαστεί οι επιβάτες. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι ε, η πρόσβαση και οι τιμίες πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε θα ευνοούν την ανάπτυξη του τουρισμού. Γνωρίζουμε ότι οι αεροπορικέ εταιρείε ήδη αξιολογούν κατά πόσον θα πρέπει να μεταφέρουν και την έδρα τους. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένη συνέπεια στον τουρισμό είναι το γεγονός ότι ε, μια σημαντική εταιρεία low cost ε, έχει ήδη ανακοινώσει αύξηση των τιμών της. Ε, ε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα, υπάρχουν κάποιες μελέτες για το θέμα αυτό. Και επίσης γνωρίζουμε ότι οι εταιρείε ε, low cost είναι πολύ σημαντικές ε, γιατί προσφέρουν πρόσβαση σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας. Τώρα, για το Λονδίνο υπάρχουν και θετικά στοιχεία. Το Λονδίνο είναι σίγουρα ένας πάρα πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός. Ε, λέγεται για 20 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, αλλά φυσικά ε, αυτό θα μπορούσε να ευνοήσει και τον τουρισμό προς το Ηνωμένο Βασίλειο ε, το Brexit. Ε, η αλήθεια είναι βέβαια ότι ε, το brand, η Ευρώπη ως brand, ως εμπορικό σήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να αυξήσουμε τους τουρίστες μας. Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, νομίζω ότι συμφωνώ απολύτως. Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν με θεωρήσεις διαβατηρίων, με διαβατήρια και ουρές στα αεροδρόμια. Ε, ίσως λοιπόν θα μπορούσε να γίνει μια αξιολόγηση και σε οικονομικούς όρους και ε, σε όρους ε, ελκυστικότητας του κάθε προορισμού. Ε, επίσης, ε, αναφέρθηκε και το θέμα της ασφάλειας. δεν είναι μόνο αυτό. Η, υγεία και η υγειονομική περίθαλψη είναι πάρα πολύ σημαντική και τα λαμβάνουν υπόψη τους οι τουρίστες για να επιλέξουν προορισμό. Επομένως αυτό θα πρέπει να προσθεθεί και στην πρακτική πτυχή που αφορά και την οδηγία που αφορά την ασφαλιστική κάλυψη. Ε, κλείνω με ένα τελευταίο επιχείρημα. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ε, πονάει αρκετούς, αφορά την ε, ε, Next Tour και αφορά το Γιβραλτέρ. Ξέρω ότι είναι ταμπού και στην Επιτροπή μας και όχι μόνον. Δεν μιλάει κανείς για το Γιβραλτάρ, ας μιλήσουμε για τη γραμμή της Κονσεψιών. Δεν αναφέρονται πουθενά αυτά όλα στα ψηφίσματα τα οποία έχουμε εγκρίνει για το Brexit, μίλησε για την Ιρλανδία, αλλά κανείς δεν μιλάει για το Γιβραλτάρ. Και νομίζω ότι αυτό είναι λάθος, γιατί σήμερα δυστυχώς υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που έχουν σταματήσει στο Συμβούλιο ακριβώς για το θέμα του Γιβραλτάρ, που κατά την άποψή μου δεν είναι δυνατό να το αποδεχτούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά νομίζω ότι έχει αφορά και το, αφορά και το θέμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, γιατί υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που ζουν στη συνοριακή γραμμή και πρέπει να πάνε στο Γιβραλτάρ για λόγους εργασίας και αύριο μπορεί να μην μπορούν να προστατεύονται καταλήλως. Επομένως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι πρέπει να το αναλάβουμε ως βουλευτές και να ασχοληθούμε και με αυτά τα θέματα και να μην ε, ε, ξεχνάμε ότι ναι μεν υπάρχουν επικρίσεις αλλά αυτοί που εκπροσωπούμε περιμένουν να τους επιλύσουμε και τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ιζαμπέλα. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσω και τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Μία ερώτηση έχω. Ίσως θα μπορούσα να την απευθύνω στον ε, Μάρκ Τάνζεν από το ΑΠΤΑ. Είπατε πολύ σύντομα, αλλά με πολύ ζωφερό τρόπο, για τον αντίκτυπο της διαταραχής ε, στην αεροπορία και τη συμφωνία για το Blue Skies, για το καθαρό ουρανό. Ε, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα περισσότερα Πού βλέπετε ότι θα κινηθούν οι διαπραγματεύσει, ε, τι δυνατότητες βλέπετε να έχουν οι Βρετανοί τουρίστες αλλά και οι Ευρωπαίοι τουρίστες ε, που πάνε στη Βρετανία και πώς θεωρείτε ότι θα ε, τους επηρεάσει οποιαδήποτε διαταραχή ε, και διακοπή τη συμφωνίας για τους ανοιχτούς ουρανού. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Συγγνώμη, θα ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις και μετά θα σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε. Ο κύριος Πίπερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Από ό,τι φαίνεται στο παράδεισο ζούμε εδώ. Όταν βλέπω τι στερείστε εσείς ε, στη, στη Βρετανία την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ε, του Open Skies, ε, θεωρήσεις, ε, το roaming, ρυθμίσεις προστασίας του καταναλωτή, τότε εμείς εδώ βρισκόμαστε σε τέλεια θέση. Και να σας ρίξω πίσω το μπαλάκι στον κύριο Τάνσερ από την Άπτα. Ε, είπατε ότι είσαστε ουδέτεροι ως προς το Brexit. Ε, γιατί, γιατί δεν είσαστε επιθετικά υπέρ του Remain, της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, εάν όχι, τότε είσαστε κι εσείς οι συνυπεύθυνοι που βρισκόμαστε εδώ σε αυτή τη θέση. Δύο συμπεράσματα. Γραμμή του προϋπολογισμού για τον τουρισμό. Δεν πιστεύω σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά σύνορα, έχουμε τη μετανάστευση, πρέπει να προωθήσουμε το Εράσμους, ε, έχουμε την έρευνα, έχουμε ένα σωρό προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε. Ε, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ γραμμή προϋπολογισμού για τον τουρισμό. Φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμπεριληφθεί στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, εσείς ασκείτε πίεση στην Βρετανική κυβέρνηση ώστε να ακολουθήσει ένα πρότυπο ε, που να προσεγγίζει όσο γίνεται την εσωτερική αγορά. Ε, πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος. Ο η κυρία Τζιλ Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας γιατί πολύ ενδιαφέρουσες, αν και καταθλιπτικές ε, παρουσιάσεις τους, όχι όμως και απρόβλεπτες, γιατί είχαμε προεξοφλήσει όλα αυτά τα αποτελέσματα σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην Επιτροπή Περιφερειών συζητήθηκε αυτό το θέμα, στην ε, διαπεριφερειακή ομάδα που θα συνεργαστεί με τις περιφέρειες προκειμένου να τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Και αυτό θα ήθελα, αν όχι σήμερα κάποια στιγμή, ε, να το αναλύσουμε. Και εγώ εκπροσωπώ την Ουαλία και κάτι που μας κάνει περήφανο στην Ουαλία είναι η εγκαρδιότητα και η φιλοξενία των Ουαλών. Ενώ στη Σκοτία δεν φαίνεται να επηρεάστηκε ο τουρισμός. Δηλαδή δεν αποκαρδιώθηκαν οι τουρίστες από την επίσκεψη στην Σκοτία και διαρωτώ με αυτό και για το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω αν μιλούσατε μόνο για το Λονδίνο ή για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρατηρήθηκε το τελευταίο χρόνο αύξηση του αριθμού των επισκεπτών των ταξιδιωτών προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Πού οφείλεται αυτό. Ίσως ήθελαν όλοι να προλάβουν να επισκεφτούν το Ηνωμένο Βασίλειο πριν το Brexit. Άρα κάτι τέτοιο δεν προϊονίστηκε πολύ θετικά στοιχεία για το μέλλον. Γιατί στις διαπραγματεύσεις για το Brexit πολλά ερωτήματα μένουν μετέωρα προς το παρόν και αναπάντητα. Οπότε δεν μπορούμε να τα καλύψουμε ούτε εδώ. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Μας έδωσαν σαφή εικόνα της κατάστασης. όσον αφορά τον τουρισμό και στην Ευρώπη αλλά και στα Βρετανικά νησιά η Μεγάλη Βρετανία μετά την πρώτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσχώρηση Πολωνίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας και των Βαλτικών χωρών Ρουμανίας, Βουλγαρίας. Ε, χρησιμοποίησε εργατικό δυναμικό από αυτές τις χώρες. Άλλες χώρες δεν το έκαναν αυτό διότι ε, είχαν προβλήματα ε, στις δικέ τους αγοράς εργασίας. Η Γερμανία, παράδειγμα, ανέβαλε ε, την ε, ελεύθερη ε, προσέλευση των ανθρώπων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτές τις χώρες εργάζονται στον τομέα παροχής υπηρεσιών στην Βρετανία. Ακούσατε τα στοιχεία, 240.000 στη Σκοτία και μόνο. Και αναρωτιέμαι, Πώς θα διασφαλιστεί αυτός ο τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Θα γίνουν διαπραγματεύσεις. για διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ε, Ευρωπαίων ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και των ε, Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, θα λειτουργήσει και στην πράξη προσβασιμότητα, ε, απαλλαγή από θεωρήσεις, ε, πώς θα λειτουργήσουν αυτά. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν ε, τόσο ενταγμένο όσο άλλες χώρες, παρόλα αυτά υπήρχε ίσχυη η ελεύθερη κυκλοφορία και ακόμα και οι επιχειρήσεις χαμηλού κόστους μπορούσαν να εργαστούν με πολύ άνεση. οι ε, διάφορες περιφέρειες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, είτε μιλάμε για τη Σκωτία είτε μιλάμε για την Ουαλία. δεν ανησυχώ πολύ για το Λονδίνο. Όταν βλέπω τις ειδήσει ε, στη Γερμανία θα πίστευε κανείς ότι ε, η βασιλική οικογένεια ε, βρισκόταν στη Γερμανία όταν ακούει για παράδειγμα για το νέο πριγκυπόπουλο της Βρετανίας. Ε, αλλά πώς θα στηρίξουμε τους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό. Ας θυμηθούμε η UKIP και άλλοι που πήραν την πρωτοβουλία για το Brexit, πώς ε, έλεγαν με μεγάλες ε, πινακίδες ότι 350 εκατομμύρια λίρες ε, σπαταλώνταν κάθε εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή τις πολιτικές εξελίξεις ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πιθανή μεταβατική ρύθμιση καθώς και ένα πιθανό νέο δημοψήφισμα. Θα δούμε. Σα Σας ευχαριστώ. Δεν ζητά άλλο ευρωβουλευτής το λόγο. Οπότε μπορώ να ξαναδώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για να απαντήσουν, να σχολιάσουν. Τόμ, χρόνου φίδου. Απλώς να επαναλάβω και θα αφήσω τις ερωτήσεις προς τον Μακ Τάνσερ για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, κυρίως που είναι ένα δίκτυο ε, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Είδαμε το έγγραφο με τις θέσεις τους και ανησυχούν για το αντίκτυπο που θα έχει το Brexit σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μαρτάντσερ, ε, θα σταθώ σε δύο ερωτήσεις που απευθύνθηκα σε μένα. Η μία αφορούσε την πολιτική αεροπορία και τους κινδύνους. Πάντως ε, ευελπιστώ ότι θα συνεχιστούν οι πτήσεις ε, ε, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να είμαστε στην ΙΑΣΕΤ, τον οργανισμό. δεν μπορούμε να έχουμε διμε... Θα μπορούσαμε να είχαμε διμερεί συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας με πολλές χώρες, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε στον οργανισμό. Αποκλείεται να συστήσουμε δικό μας οργανισμό. Δεν υπάρχει καν τέτοιο ενδεχόμενο, ούτε ω σε διεκτάκτο ανάγκης. Ε, πάντως, ε, ακόμη και γίνει κάτι θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις ε, και μέχρι να συστηθεί θα υπάρχει δυναμία πραγματοποίηση πτήσεων. Οπότε το θέμα αυτό πρέπει να διευθυνθεί κατεπηγόντως. Σε ό,τι αφορά την ουδετερότητά μας ε, στο δημοψήφισμα, όταν κάναμε την ανάλυση μας για το πόσο επιζήμεθα είναι για τον τουρισμό, το επισημάναμε στον κόσμο με διαβήματα προ τα ΜΕ. Και για τον τουρισμό είδαμε περισσότερες αρνητικές παραθετικές συνέπειες. Βέβαια ήταν κάπως συγκεχημένα τα πράγματα και λίγο αρπακόλα. Πάντως η πραγματικότητα είναι ότι αν πά στον κόσμο και τους πει πώς να ψηφίσουν, ε, θα δημιουργήσει αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτέλεσματα. Ενώ αν ε, ε τους δώσει επιχειρήματα για το πώς θα επηρεαστεί η καθημερινότητά τους, τότε θα κάνουν μόνοι, μόνοι τους τις επιλογές τους. Πάντω για τι επιχειρήσει ε, για ένα θέμα που είναι τόσο συγκινησιακά φορτισμένο και το ευαίσθητο, αν κανεί ε, πάρει έντονα το μέρο μια πλευρά, κινδυνεύει να χάσει του μίσου πελάτε του. Και μάλιστα τι στιγμέ του δημοψηφίσματο και επιχειρήσει και επαγγελματικέ και εμπορικές οργανώσεις ε, ήταν πολύ προσεκτικές. Πάντως ε, επισημάναμε τι δυνητικέ αρνητικέ συνέπειε του Brexit και πριν το δημοψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ θα σχολιάσω δύο ερωτήσεις. Η μία της κυρίας Δεμόντε για το, το Γιβραλτάρ. Το Γιβραλτάρ δεν είναι ταμπού. Έχει ειδικό καθεστώς γιατί πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι 13.251 αυτοί οι, παρα, οι μεθοριακοί εργαζόμενοι και δεν ξέρω αν είναι του θέματος. Ε, και δεν ξέρω αν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως αποσπασμένοι ή ε, διαμεθοριακά εργαζόμενοι. Πάντως ε, είναι θέμα της δημόσιας συζήτησης. Εγώ ε, αυτό έχω να πω για το Γιβραλτάρ. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Evans για το πώς λειτουργεί η διαπεριφερειακή ομάδα για το Brexit στην Επιτροπή των Περιφερειών, πρόσφατα συστήθηκε πριν τρεις-τέσσερις εβδομάδες αυτή η διαπεριφερειακή ομάδα Καθορίστηκαν τρεις άξονες ε, εργασίας. Πρώτα, ανταλλαγή πληροφοριών για τις πιθανές συνέπειες του Brexit. Δεύτερος άξονας, πολύ σημαντικός των εργασιών, ε, εντοπισμό των περιφερειών που θα πληγούν περισσότερο ή που είναι πιθανό να επηρεαστούν ιδιαίτερα από τις συνέπειες του Brexit και συνεργασία με τις περιφέρειες αυτές για να δούμε πώς μπορούμε να μετριάσουμε τις επιζήμιες συνέπειες του Brexit. Και τρίτος άξονας αφορά το μέλλον. Ε, θα πρέπει με τις περιφέρειες με τις οποίες συνεργαζόμαστε να αναπτύξουμε κάποιες ιδέες για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας αυτή και στο μέλλον. Αυτή η διακομματική ομάδα ε, προεδρεύεται από τον κύριο Τεκώστερ από τη Γαλλία και έχει δύο αντιπροέδρους. Ο ένα είναι από τις κατοχώρες και ο δεύτερος από την Ιρλανδία. Η επόμενη συνεδρίαση αυτής της ε, διακομματικής ομάδας ε, δεν ξέρω πότε θα είναι, πάντως θα συνεδριάζει περίπου 7-8 φορές το χρόνο. Ευχαριστώ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Πάντως, στο μέτρο που αρχίζει και ο κλάδος να εγκύπτει στις επιπτώσεις, καλό είναι να συγκεντρώνουμε όλα τα στοιχεία και να συμπληρώνουμε το τοπίο, γιατί στο μεταξύ θα διευκρινιστούν κάποιοι προς το παρόν άγνωστοι οι αστάθμητοι παράγοντες, οι απρόβλεπτες συνέπειες. Κάποιος ανέφερε την ασφάλεια υγείας ή ασφάλεια αυτοκινήτου, χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σίγουρα θα έχουμε επιπτώσει σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Θα πρέπει να εντοπίσουμε τα θέματα αυτά και να τα αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά στο μέτρο που ανακύπτουν. Και ο Νάιτζελ Μόργαν, σε ό,τι φορά τις ερωτήσεις, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν καταρτιστεί μεγάλες εμβέλειας μελέτες για τον αντίκτυπο που θα έχει το Brexit ε, στις αεροπορικές μεταφορές, της στους αερομεταφορείς. Δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε, ούτε υπάρχει και σαφήνεια από την κυβέρνηση, αλλά δεν υπάρχει καν ε, αντίληψη σαφής ε, για τις συνέπειες του Brexit στον τουρισμό γενικώ. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στην φιλοξενία, δεν έχουμε τέτοιες έρευνες και οι περισσότερες πληροφορίες ε, είναι αποσπασματικές και έχουν λουθεί από συγκεκριμένε οργανώσεις. Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει ε, πλήγμα στην ε, τουριστική φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου. Για πολλούς Ευρωπαίους ακόμη θεωρείται φιλόξενος προορισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι ελλειπείς οι πληροφορίες που έχουμε και στο ερώτημά σας για το Λονδίνο. Από τη σκοπιά της Ουαλίας και φαντάζομαι και ο Μάλκορ θα το έλεγε από τη σκοπιά της Σκοτίας είναι τεράστια η πρόκληση των περιφερειών και άλλων χωρών της του Ηνωμένου Βασιλείου, το άλλο του Ηνωμένου Βασιλείου να προσελκύσουν ε, τουρίστες και να τους αποσπάσουν από το Λονδίνο που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο τουριστών. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό. Και τώρα, αν θα συνεχιστεί και σε τι βαθμό, τι να σας πω, δεν το γνωρίζω. Πάντως, το δικό μου μήνυμα θα ήταν ότι θέλουμε μεγαλύτερη σαφήνεια για τα επιχειρησιακά θέματα, για όλα τα επιμέρους ζητήματα που επισήμανε οι συνάδελφοι και χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση και πιο συγκεκριμένες έρευνες για τα θεμελιώδη ζητήματα και τις βασικές συνέπειες τους. Ευχαριστώ Νάιτζελ. Οπότε θα ήθελα να διαρωτηθούμε, συνάδελφοι. Ποια είναι τα συμπεράσματα της ακρόασης αυτής. Δεν μ' αρέσουν ε, οι συνεδριάσεις ε, με μακροσκελέστατες συζητήσεις αλλά καμία συνέχεια. Οπότε θα έκανα την εξής πρόταση να συγκεντρώσουμε τις ομιλίες σας, ε, τα σχόλιά σας, ε, τα PowerPoint που παρουσιάσατε και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και να τα στείλουμε στους ηθήνοντες ε, της πολιτικής. Γιατί αυτή ήταν μόνο μια συνεδρίαση της ειδικής ομάδας τουρισμού της Επιτροπής Μεταφορών, αλλά καλό θα ήταν να προβάλλουμε γενικότερα αυτές τις απόψεις. Θα στείλω λοιπόν το υλικό σε όλους τους ευρωβουλευτές αλλά και στις κυβερνήσεις, στη Βρετανική κυβέρνηση και στους αξιωματούχους εδώ των Βρυξελών. Αν μπορούμε να το κάνουμε σύντομα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, γιατί πραγματικά ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα σε αυτή τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και ελπίζω να ήταν χρήσιμη για όλους αυτή η συζήτηση και κυρίως το πέρας της ε, συνεδρίασης της Επιτροπής. Ραντεβού την επόμενη φορά στις 14 Μαΐου, 3 το απόγευμα. Γεια σας.